guten Tag. Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε τις συνεδρίες παρακαλώ. Έχει κανείς για την ημερήσια διάταξη. Ουδής. Πολύ καλά. Δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης έγκριση των πρακτικών της περασμένης συνεδρίασης. Αν έχετε κάτι να πείτε για τα πρακτικά, πείτε τα μου μέχρι το τέλος της μέρας, αλλιώς θα τα θεωρήσω εγκεκριμένα. Υπά... Σήμερα ε, έχουμε web streaming στη συνεδρίαση, άρα πρέπει να έχουμε κοσμία συμπεριφορά όλοι μας. Όσον αφορά τη διαρμηνία υπάρχουν σωρό γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Ε, Ολλανδικά μπορεί κανείς να ακούσει, να μιλήσει αλλά δεν μπορεί να ακούσει. Επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, το σημείο 4, οι πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση της UNESCO 2005 και η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρονται στην πολιτιστική ποικιλομορφία η οποία θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να περιλαμβάνεται με κάποια έννοια σε όλες τις πολιτικές. Οι εξωτερικές υπηρεσίες της... Can I ask you to be a little bit uh, quiet, Λίγη ησυχία ζητάει η κυρία Πάκ στην αίθουσα. Λοιπόν, είναι η σωστή στιγμή λοιπόν να συζητήσουμε τις πολιτιστικές διαστάσεις στις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να εκπονήσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε η κυρία Σάκε. Στις 12 όχι, στις 9 Δεκεμβρίου είναι η ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Αν όμως σήμερα μετά από τη συζήτηση που θα κάνουμε καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες, τότε θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Διότι Δεν ε, είναι πήγοντα τα θέματα. Ε, μπορούμε να τα αφήσουμε για το Γενάρη. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην κυρία Σάκε, η οποία θα μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Μαρίκε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, mm. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη έκανες και τόσο φροντισμένη εισαγωγή για το θέμα και να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους, ε, Επιτροπή, Συμβούλιο, μη κυβερνητικέ και του άλλου εμπλεκόμενου που συμμετέσχουν σε αυτό το πρώτο σχέδιο κειμένου ότι του ευχαριστώ για τη συμβολή του, διότι πρόκειται πραγματικά για ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, το οποίο θα κάνει τώρα τη διαφορά που έχουμε συγκροτήσει στην εξωτερική υπηρεσία. Βέβαια, από την άλλη μεριά, συγκεκριμένε προτάσει δεν έχουν κατέβει σε σχέση με το τι θα γίνει με τον πολιτισμό που για μας αυτό δικαίως είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τις πολιτικές Ευρωπαϊκές Ένωσης, για την ταυτότητα, για την ε, πολυμορφία. Όμως το ερώτημα είναι πώς μπορεί να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια ούτω ώστε να εντάξουμε την πολιτική, να κάνουμε το mainstream σε όλες τις πολιτικές που ασκούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά τον προϋπολογισμό, με δεδομένο ότι τα ε, προγράμματα του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είμαστε στην ευτυχή θέση να μην χρειάζεται να ρωτήσουμε περισσότερα χρήματα, απλώς να γίνουμε πιο στρατηγικοί, πιο αποτελεσματικοί για τα προγράμματα που ήδη τρέχουν και για τους πόρους που ήδη ε, έχουν ε, παρασχεθεί. Για να δούμε τώρα μερικά σημεία από την, Ευρωπαϊκή, από την έκθεση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καλύψουμε όλα όσα θα θέλαμε να καλυφθούν στο πρώτο σχέδιο κειμένου και για αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχαμε τόσους που βοήθησαν γιατί έτσι η έκθεση γίνεται πιο συγκεκριμένη, πιο πλήρης όπου χρειάζεται. Τώρα σε σχέση με τα πολιτικά προγράμματα και τις πολιτικές μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση. Δύο είναι οι τόποι που διαδραματίζει κάποιο ρόλο ο πολιτισμό, τα προγράμματα που συζητούμε εμεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, media, ε, παιδεία, κληρονομιά, τα αεραστεχνικά, όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με ταυτότητα, τέχνες ε, και ασχολούνται με αυτά άμεσα. Μια άλλη μεριά, ο πολιτισμός και τα πολιτιστικά χρησιμοποιούνται όλο ένα περισσότερο και θεωρούνται περισσότερο ως ένα μέσο. Μέσο για να ε, συσφίξουν τις σχέσεις μας με τους λαούς άλλων χωρών και να συμφιλώσουν μετά από κάποιες συγκρούσεις ε, τους λαούς ή το να βοηθήσουμε την ανάπτυξη ανθρώπινα δικαιώματα, ε, τη συμμετοχική δημοκρατία και όλα αυτά δεν είναι μόνο προγράμματα που ε, έχουν ως πλατφόρμα και θεμέλιο κάποιες αξίες, αλλά έχουν να κάνουν και με την αναβάθμιση των οικονομικών δυνατήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αναβάθμισης των εξωτερικών σχέσεων με την εγκατάσταση επιχειρήσεων, τουρισμό, Επομένω είναι ευκαιρία που δεν μπορούμε παρά να την λάβουμε υπόψη. Όπω προείπα, προ το παρόν έχουμε κάποια προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με τι πολιτικέ σχέσει. Ακόμα έχουμε εδώ μια κατάτμιση σημαντική σε σχέση με τι διάφορε πολιτικέ τη Ένωση. Α πούμε, έχουμε και πόρου για τον πολιτισμό και κονδύλια τα οποία έχουν δεσμευθεί. Ε, σε σχέση με τι εταιρικέ σχέσει, χώρες ΑΚΕ, γειτονική σχέση, εταιρική σχέση με, την Ανατολία, αλλά επίση και με συντονισμένη στρατηγική πολιτική και επομένως και εμεί ε, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μα σε όλα αυτά και βέβαια εμεί εδώ ξέρουμε τι πάνε πει και πόσο αξίζει ένα πολιτικό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να σα πω ότι στην έκθεση τονίζω το ρόλο τη Ευρωπα... της ε, υπηρεσίας δράσεις. Και εκεί θα πρέπει να περάσει το μήνυμα. Και είναι ηρωνικό το ότι καμιά φορά ε, αυτό δεν γίνεται τόσο, τόσο εύκολα αντιληπτό. Ενώ τι γίνεται στον πολιτισμένο κόσμο μας, η Κίνα, άλλη παίκτεση, η ΙΠΑ, ακόμα και το ΝΑΤΟ, όλα ένα και περισσότερο χρησιμοποιούν προγράμματα πολιτιστικά, πολιτιστική διπλωματία, επίσης και σε σχέση με την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδυασμό με τα αντίστοιχα προγράμματα. Ούτω ώστε να διαδώσουν αυτές τις ε, αξίες, οπότε και εμείς να μην χάσουμε το τρένο, να είμαστε και εμείς ένας παγκοσμίο παίκτη παρά το ότι θα πρέπει και εμείς να ενεργήσουμε ως τέτοιος παίκτη να δούμε τις άρεστες πρακτικές των κρατομελών να τις χρησιμοποιήσουμε, μην να φεύγουμε τον τροχό απλώς, να τις χρησιμοποιήσουμε τις αυτές τις άρεστες πρακτικές, να τις συντονίσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε μία ομογενοποιημένη ευρωπαϊκή κουλτούρα και πολιτισμό, αλλά θα είναι αυτός ο πλούτος της πολυμορφίας που θα αξιοποιείται όσο γίνεται καλύτερα. Ή στα θέματα δε που εμείς εδώ συζητούμε, αλλά και γενικότερα διαπιστώνεται ότι έχουμε κάποια νέα μίντια, νέα μέσα που έχουν αυξανόμενη σημασία για τα πολιτιστικά και είναι μια άριστη ευκαιρία ούτως ώστε κανείς να μοιραστεί αυτό το περιεχόμενο του πολιτισμού και από απόσταση και να δούμε πώς είναι δυνατόν όλα αυτά θα διευκολυνθούν με το, με το και με άλλους τρόπους. Να δούμε επίσης πώς η ψηφιακή τεχνολογία έχει σχέση με τα πολιτικά προγράμματα και επομένως Νομίζω ότι θέλουμε πιο συνεπή, πιο συνεκτική πολιτική, ούτω ώστε να έχουμε πολύμορφα διαφορετικά προγράμματα όπως τα χρησιμοποιούμε και για να βοηθήσουμε την υπόθεση της δημοκρατίας και ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ό,τι θέλετε πέστε μου και ευχαρίστως τις σκέψεις σας να τις καλύψω στη επόμενη φάση της Ευχαριστούμε πολύ, λέει η πρόεδρος. Μέχρι στιγμής δεν ζήτησε κανείς το λόγο, αλλά τον ζητώ εγώ. Λοιπόν. Ich habe ein Problem. Έχω ένα πρόβλημα. Το... που σχετίζεται ίσως <laughs> και με τον εισηγητή. Ο εισηγητής αγαπάει ιδιαίτερα το διαδίκτυο και την ψηφιακή εποχή. Αλλά ακόμη και στην ψηφιακή εποχή υπάρχουν και άλλα οπτικοακουστικά μέσα. Καινούρια. Αντί για ίντερνετ λοιπόν θα πρέπει στην έκθεση να έχουμε έναν όρο που περιλαμβάνει και άλλα ε, μέσα. Επίσης το σημείο 20 που έχει στην έκθεση όπου ζητάς η Επιτροπή να ενεργοποιηθεί και να εγκρίνει μια πράσινη βίβλο δεν διαφωνώ αλλά νομίζω ότι αντιθέτως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της έκθεσης οπότε πρέπει να μπει σε πιο κυριαρχή και προφανή θέση μετά μιλάς για digital diplomacy, ψηφιακή διπλωματία. Για μένα θα έπρεπε να μιλάς για digital, για cooperation, συνεργασία. Και στο 13 που έχει τον όρο global paper, player, παγκόσμιος παράγοντας, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να μιλούμε για global responsibility, ευθύνη, παγκόσμια ευθύνη. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε και να προβάλλουμε περισσότερο την ε, σύμβαση της UNESCO που ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η, ε, τα κράτη-μέλη την εφαρμόζουν σωστά όλα αυτά που καταφέραμε αποδυναμώνονται από την πίσω πόρτα. Και τούτη εδώ η έκθεση, ε, αν δεν προβάλλει αυτό, αυτή τη σύμβαση, θα παίξει το παιχνίδι αυτών που θέλουν πραγματικά να αποδυναμώσουν τη σύμβαση της UNESCO. Ενώ εμείς αγωνιστήκαμε για αυτήν. Αυτά λοιπόν σαν πρώτες παρατηρήσεις ε, από πλευρά μου που θα ήθελα να προσέξει η Μαρίκε. Α, και κάτι τι άλλο. Δεν θα ήθελα να μιλάς συνέχεια για προγράμματα, διότι δεν πρόκειται για προγράμματα, πρόκειται για δράσεις. Action. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε λοιπόν να κινούμεθα στο ίδιο μήκος κύματος και αυτό ίσως να διευκολύνει και τη συζήτηση. Ο κύριος Φλέκενστάιν. Ναι κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή, μάλλον την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης αυτό. Ευχαριστώ και σας Πρόεδρε για τις παρατηρήσεις που μόλις τώρα κάνατε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για το σημείο 20 όπως κάνατε και εσείς και να πάω ένα βήμα πιο πέρα. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια αν θέλουμε πραγματικά να φτιάξουμε μια στρατηγική, ένα concept όπως λέμε. Είναι σωστό αυτό να το αναθέσουμε στην Επιτροπή, στην Κομισιόν. Μήπως θα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάποιες πρώτες σκέψεις για τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής στρατηγικής. Να, ε, να μιλήσουμε, να δούμε ποια είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να καλύπτει μια τέτοια στρατηγική. Δεύτερη παρατήρηση. Ήδη Υπάρχουν δραστηριότητες, προγράμματα, πρωτοβουλίες και στην, ε, στις εξωτερικές δράσεις, στην εξωτερική δράση που περιλαμβάνουν και την κουλτούρα, τον πολιτισμό. Εδώ πρόκειται για την εμείς θέλουμε απλώς να κάνουμε κάτι πέρα από τη διαχωριστική γραμμή και από αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη στον τομέα των εξωτερικών δράσεων. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο που θα ήθελα να, να τονίσω. Το σημείο 11 όπου ζητείται η μεταρρύθμιση του ορισμένων πραγμάτων. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι γιατί θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοεί η κυρία Σάκε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αναδιατυπώσουμε το 11. Επίσης θα ήθελα να κυρία Πρόεδρε, να συμφωνήσω με αυτό που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε το, το θέμα δεν είναι τόσο επίγον οπότε δεν πρέπει με κάθε ε, για κάθε λόγο να για κανένα λόγο να βιαστούμε ή και οι συγγήτρια και οι σκιώδεις θα πρέπει να καθίσουν να ξεβεδιάσουν τα θέματα και να πάμε ίσως λίγο πιο αργά. Ευχαριστώ πολύ λέει η πρόεδρος ο κύριος Κάβαρεκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Μαρίζα Σάλκε και για την τόσο καλή δουλειά που έκανε στο συντονισμό της, των διαφόρων προσεγγίσεων που είχε ο καθένας μας σε αυτό το φάκελο. Είχαμε πολλές ανταλλαγές απόψεων και βλέπουμε πολύ συχνά ότι η δουλειά της είναι πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου σε, ένα, σε μια πτυχή που θεωρώ ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω στην έκθεση και με απασχολεί οφείλω να ομολογήσω. Παραδοσιακά νομίζω ο πολιτιστικός παράγοντας ε, στις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και γενναίες ολόκληρες, ήταν μία μονάδα, αν θέλετε, πολιτιστικών εξαγωγών προς τα 27 κράτη-μέλη χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις δηλαδή σαν ένα μέσον για να εξάγει την ταυτότητα του κράτους, δηλαδή την γαλλική, την πορτογαλική ταυτότητα κτλ. Η ισπανική λογοτεχνική παράδοση, η γερμανική λογοτεχνική παράδοση κτλ. Μέσω των υπηρεσιών που γνωρίζουμε, το Ινστιτούτο Θερβάντες, το Ινστιτούτο Καμόες, το Ινστιτούτο Γκέτε κτλ. Έχουμε την ευκαιρία με την ε, υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουμε κάτι παραπάνω και να ξεπεράσουμε, αν θέλετε, αυτόν τον πολιτιστικό ακόλουθο στα, στις διπλωματικές υπηρεσίες. Και δεν, δεν θα ε, λειτουργεί απλώς και μόνο σαν ε, εξαγωγέας, η, αυτός ο η πολιτιστική πτυχή θα είναι και εισαγωγέ, θα μπορούμε, θα μπορούμε να κάνουμε και εισαγωγέ και εξαγωγέ αν θέλετε. Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, την Ευρώπη δεν πρέπει να τη δούμε μόνο σαν έναν ε, σφαιρικό παράγοντα, αλλά σαν ένα παράγοντα με σφαιρικές ε, ε αρμοδιότητες, ένα παγκόσμιο παράγοντα. Δηλαδή, Είμαστε ένας παγκόσμιος παράγοντας, ο οποίος όμως μπορεί να ε, δέχεται και επιρροές από όλο τον κόσμο. Αυτό κάνει πλούσια την, την Ευρώπη. Δηλαδή, το άτομο το οποίο θα, είναι σαν, θα λειτουργεί σαν κεραία στις ε, διάφορες αντιπροσωπείες μας στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος όχι μόνο θα διαδίδει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά θα πρέπει να δέχεται και όλος έχει να προσφέρει ο κόσμος, ο υπόλοιπος κόσμος. Μιλάω θεωρητικά αυτή τη στιγμή, αλλά όλοι ξέρετε τι θέλω ακριβώς και προς τα που πηγαίνω. Πρέπει να δώσουμε δηλαδή μια πολιτιστική διάσταση στις, ε, στον εξωτερικό τομέα και να λειτουργήσουμε ε, με καινοτόμες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Δυστυχώς, α, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ακόμη παρατήρηση. Από τη μια μεριά ε, χαιρετίζω αυτό που έκανε η συγγήτρια, γιατί και εγώ Μα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ίντερνετ, ε, υποστηρίζω αυτό που λέει, όμως βεβαίως μια και μιλάμε εδώ για πολιτιστική ποικιλομορφία και τα λοιπά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και άλλα μέσα και άλλα εργαλεία και άλλες, ε, άλλους τρόπους. Δεν είναι μόνο με το ίντερνετ που θα ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον γύρο κόσμο. Το, Κάτι άλλο όμως θα ήθελα να πω είναι το εξή. Είναι γεγονός ότι μια κοινή εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί κάλλιστα να προβάλλει προς τα έξω τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία της Ευρώπης. Όμως υπάρχει και η πολιτιστική ποικιλομορφία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί και οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες προβάλλουν τις δικές τους ε, κουλτούρες και παραδόσεις προς τα έξω η κοινή πολιτιστική η κοινή κουλτούρα της Ευρώπης πρέπει να προβληθεί αλλά να τονιστεί ιδιαίτερα και αυτό που εμπλουτίζει την Ευρώπη ε, η ιδιαιτερότητε διαφόρων κρατών μερών. σε θέματα πολιτισμού. Πρέπει να τονιστεί και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Πακ. Να προσθέσω δύο πράγματα. Στο σημείο 28 λέει ζητεί τη χάραξη μιας στρατηγικής για την προαγωγή των ευρωπαϊκών πολιτισμικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Θα μπορούσαμε εδώ να βάλουμε αυτό που ζητεί ο κύριος Φλάκενστάιν. Δηλαδή να βάλουμε συγκεκριμένους στόχους και, ε, και πιο συγκεκριμένα πράγματα για δηλαδή το πού μπορούν να γίνουν αυτά. Ε, το, δεν ξέρω αν θυμάστε την Όινικ, την Όινικ που ήρθε εδώ και μας επισκέφτηκε που είναι ουσιαστικά Bridge Council, Cervantes, Goethe Institute, Alliance Française και Institut Français κτλ. Αυτοί ενώνονται στην UNIC και είναι πρόθυμοι να κάνουν ορισμένα πράγματα σαν Ευρωπαίοι με στα πλαίσια της ΕΝΙΚ. Τονίζω λοιπόν αυτό που είπαν οι συνάδελφοι και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λιγάκι το 28 Τώρα στο 5 εκεί που λέμε ότι θεωρεί σημαντική τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τις πολιτιστικές πτυχές εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όμως φαίνεται να ξεχάσατε αγαπητέ, αγαπητοί συνάδελφοι την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να βάλουμε εδώ και την κοινωνία των πολιτών. Κατά τα άλλα η έκθεσή σα είναι μια καλή βάση για συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί λίγο και να αναδιατυπωθεί ούτω ώστε να τονιστούν οι στόχοι και όπως είπε ο κύριος Φλέγκεστάιν, να μπορούμε να υποδείξουμε στην Κομισιόν προς τα που θέλουμε να πορευθούμε. Και εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα, αλλά δίκιο έχει ο Φλέγκεστάιν που λέει ότι δεν μπορούμε να τα αναθέσουμε όλα στην Κομισιόν, να καθίσουμε και εμεί να σκεφτούμε μερικά πράγματα, να κάνουμε κάποιε υποδείξει ώστε να ξέρει πού θα που, προς τα που θέλει να πάει. Και τώρα θα δώσω το λόγο ακριβώς στην Κομισιόν. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Πρώτα-πρώτα σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία μας δίνετε να εκθέσουμε τις αρχές μας σκέψεις σε αυτή τη φάση. Τρία Τι να σας πω που είναι τα βασικότερα. Πρώτα Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτό το κείμενο που η έχει συντάξει Όσον αφορά την γενική μας διεύθυνση και εμείς ε, συμφωνούμε με την ανάλυση ε, για την μέχρι εδώ πρόοδο. Ανατρέχοντας πίσω στο 2007, τότε που εγκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Ατζέντα, ε, σίγουρα έχει συμμεθεί η πρόοδος και τα λέει κατά η έκθεση. Αυτό το καλοκαίρι πρόκειται να εγκριθεί το σχετικό κείμενο, οπότε σωστά αναφέρεται η έκθεση σε κάποιες προτάσεις για τρίτες χώρες, για ανάπτυξη δυνατοτήτων και, ότι και εμείς διαφορεμαστε πάρα πολύ στο να επενδύσουμε πάνω σε αυτές τις προσπάθειες. Επίσης, συμβαίνουν πάρα πολύ όσον αφορά την ανάλυση των προκλήσεων, γιατί ακόμα έχουμε πολλές προκλήσεις και τα λέει η έκθεση όσον αφορά το περιθώριο που υπάρχει για μελλοντική συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων θεσμικών οργάνων, κοινωνίας και λέει, αναφέρεται εδώ πέρα η κατάτιμηση των μέσων, ε, αυτό είναι κλασική εκδήλωση που αφορά τέτοιες προσπάθειες. Επίσης, έχουμε την πρόταση για τα μελλοντικά προγράμματα. Ό,τι θα κάνουμε τα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Τέλος, να σας πω όσον αφορά για τα συμπεράσματα για αυτό το ευρωπαϊκό σήμα. Σήμα, μάρκα, μάλλον ε, ταυτότητα ευρωπαϊκή, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διευνήσει αυτή τη δυνατότητα. Και βέβαια ακούσαμε σήμερα ότι ο καθένας έχει διαφορετική άποψη, πολύμορφη Ευρώπη, υπεύθυνη Ευρώπη και όλα αυτά πάρα πολύ ενδιαφέροντα για προγράμματα, για πρωτοβουλίε. Και όταν λέμε για ταυτότητα ευρωπαϊκή, όχι με τίποτα εις των εθνικών ταυτοτήτων. Πολύ σωστά και η κυρία Πάκ τόνισε την συνεργασία που ήδη έχει ξεκινήσει με τα εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα, UNIC. Ευχαριστώ. Μετά την παρέμβαση των συναδέλφων δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να συμπληρώσω εγώ. Είμαι υπεύθυνο για την οπτικοακουστική πολιτική. Χαίρομαι για αυτά που λέτε και το ρόλο που λέτε ότι μπορεί να παίξει η οπτικοακουστική πολιτική. Αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω φέρω ένα, για να σας δείξω ότι κάνουμε και εμείς προσπάθειες για να ενισχύσουμε την εξωτερική πτυχή των οπτικοακουστικών. Ε, υπάρχει ένα έγγραφο ε, staff paper το οποίο φτιάξαμε πέρσι και το οποίο πραγματικά περιγράφει την πολιτική μας και ε, η οποία περιλαμβάνει και μια εξωτερική πτυχή και περιγράφεται στο έγγραφο αυτό τι γίνεται στις σχέσεις μας και με άλλους εταίρους, με τι να σας πω, με αδελφά προγράμματα, το όπως το πρόγραμμα Media ή αντίστοιχα της UNESCO κτλ. Wenn ich äh, mir die Punkte 17 17, 20, 22, 23, 24. Αν κοιτάξουμε αυτά τα σημεία, λέει η κυρία Πακ, νομίζω ότι αυτά θα μπορούσαμε να συμπτύξουμε Μαρίκα, Μαρίκε και να το κάνουμε πιο ο, συνεκτικά. Γιατί τελικά δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν ένα τροποποιηθούν μία προς μία η παράγραφη που έχει στο κείμενο μπορείς να ακούσει τα σχόλια και να συμπτύξεις ενδεχομένω σε κάποιους παραγράφους. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα τόσο χρήσιμα σχόλια. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά. Όντως ήταν μια πρόκληση να τα λάβουμε όλα υπόψη μας. Όσο περισσότερο συνοψίζουμε τόσο καλύτερα πιστεύω θα είναι τα πράγματα. Συμφωνώ ότι η συνθήκη της UNESCO πρέπει να είναι ακρογωνιαίος λίθος και θα πρέπει να εφαρμοστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλες τις χώρες. Ε, προφανώς δεν μιλάμε για προγράμματα, μιλάμε για ενέργειες, για δράσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερες δράσεις στον τομέα αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. και η πολιτιστική διαφοροποίηση, αν θέλετε, οι πολιτιστικές διαφορές νομίζω ότι ενδυναμώνουν και ενισχύουν ε, την ευρωπαϊκή πολιτιστική διάσταση και την αναφέρουμε την UNIC σαν πολύ καλή εμπειρία και θέλουμε τη συνεργασία μαζί τους γιατί δείχνουμε ακριβώς ε, πώς μπορεί να λειτουργήσει η συνεργασία κάποιων οργανισμών, οργάνων που προέρχονται από, την, ε, από τον κόσμο τέλος πάντων. Τώρα όσον αφορά τις συνεργασίες, ο κύριος Φλέκενστάιν έκανε μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερα για, για τις ιδέες σας για την μεταρρύθμιση του UPR. Ε, δεν είναι δεν είναι ότι αγαπάω ιδιαίτερα το ίντερνετ, ε, αλλά απλώς ε, για να αναγνωρίσω την πρόοδο που έχει γίνει. Οι νέοι είναι κυρίως που μπορούν να μοιραστούν ε, πληροφορίες σε μεγάλη απόσταση, χωρίς να προκαλέσουν οποιαδήποτε μόλυνση της ατμόσφαιρας ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, προφανώς υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες τις οποίες θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε εδώ και θα πρέπει να είμαστε συνετοί και δημιουργικοί όταν να τις χρησιμοποιούμε βέβαια. Τώρα, η πλευρά της αμοιβαιότητας των επαφών και οι επαφές με τις τρίτες χώρες σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όντως πρέπει να είναι αμφίδρομη η επικοινωνία με, την, με τον κόσμο, με τους πολίτες, με την κοινωνία των πολιτών σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Φερχάιεν δεν έχουμε κανένα στόχο, κανένα σκοπό να ε, επιβάλλουμε, αν θέλετε, το ψηφιακό κόσμο, αλλά ίσα ίσα να το χρησιμοποιήσουμε για να μοιραστούμε τον πολιτιστικό πλούτο που υπάρχει στην Ευρώπη. Προφανώς εδώ υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συνεισφορά τους όσον αφορά την δημιουργία δυναμικού, αν θέλετε, και της κοινωνίας των πολιτών και την UNESCO. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε ενέργειες, διότι το θέμα μας δεν είναι απλώς να χρησιμοποιούμε ωραία λόγια, αλλά να κάνουμε και κάτι το, για τις πολιτικές της οπτικο, στον τομέα θα ήθελα να ζητήσουμε ε, για να τη συμπεριλάβουμε περισσότερο. Τέλος πάντων, το κείμενο θα μπορούσε σίγουρα να είναι πιο συγκεκριμένο σε κάποια του σημεία και όταν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, και τώρα πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα. Αν παραμείνουμε στη 12η Δεκεμβρίου σαν ημερομηνία κατάθεση των τροπολογιών, μπορούμε να ψηφίσουμε το Γενάρη. Αν αναβάλουμε τη, την, ε, την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, τότε θα πρέπει να ψηφίσουμε το Μάρτιο. Για το Φλεβάρι δεν έχουμε συνεδρίαση. Φλέκενστάιν. Εδώ τα βγάλαμε πέρα τόσο καιρό δίχως μια τέτοια έκθεση. Δεν πειράζει να αργήσουμε και ένα μήνα. Άρα ας μην βιαστούμε για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Βλέπω ότι πολλοί γνέφουν θετικά, λέει η κυρία Πάκο. Πότε? 20 Λοιπόν, Η 20 Ιανουαρίου η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών και μετά ψηφίζουμε στις 3 Μαρτίου. Εν τω μεταξύ όμως θα ανταλλάξουμε απόψεις με την εισηγήτρια. Όλοι οι σκιώδες παρακαλώ να προσπαθήσουν να κάνουν προτάσεις για να βελτιώσουμε όλοι μαζί την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σάκε. Καλή δουλειά και προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που λέει η Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την υποστήριξη στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ε, 2020. Συγχωρείτε. Η συγγήτρια Μαρία Βαντία Ικουτσέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται έχουμε αλλαγές στο κοινό προσέλευσης αποχωρήσεις. Η Επιτροπή Γενικών Υποθέσεων και Απασχόληση είναι κυρίω αρμόδια επιτροπή και προσπαθούμε τώρα να δώσουμε μια όθηση στη σύνδεση του πολιτισμού με, με τα θέματα τη κατάρτιση, στα πλαίσια τη πολιτική του 2020 και όλοι οι συναρμόδιοι δουλέψαμε σκληρά για τη στρατηγική για το 2020 και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση και η παιδεία ούτω ώστε να πετύχει αυτή η στρατηγική και από δική μας πλευράς, για τη δική μας αρμοδιότητα, θέλουμε να τονίσουμε στις λεπτομέρειές τους τα σημεία εκείνα τα οποία από πλευρά παιδείας και επαγγελματική κατάρτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όπως γνωρίζετε, ε, μια τέτοια γνωμοδότηση ε, ε, έχει, έχει αυστηρή περιχαράκωση, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μακροσκελής και όπως μπορείτε να δείτε στο σχέδιο του κειμένου το οποίο σας έχω μοιράσει τα θέματα που θεωρούν τα πιο σημαντικά πρώτα πρώτα. Εδώ αναφέρω ότι στη νέα ψηφιακή οικονομία η δημιουργικότητα και οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών δημιουργούν μια νέα επιχειρηματική νοοτροπία που στενά είναι συνδεδεμένη με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Γι' αυτό θεωρώ ότι η παιδεία και η κατάρτιση θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην πολιτική μας ατζέντα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για τη στρατηγική του 2020 επίσης όσον αφορά την επένδυση σε παιδεία κατάρτιση αυτό είναι κάτι που είναι απαραίτητο για καλύτερο μέλλον της Ευρώπης. Οι δε βασικές ικανότητες και οι νέες δεξιότητες είναι οι νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους. Η βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και κατά της ε, ανεργίας. Επίσης λέμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ βασικό να βελτιώσουμε τη σχέση, τη σχέση μεταξύ ε, ιδρυμάτων και επαγγελματική κατάρτιση, γιατί έχουν γίνει εδώ κάποιε αλλαγέ όσον αφορά την ε, προετοιμασία, κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται επομένω εδώ δημιουργικότητα, να δοθεί μια όθηση, να ληφθεί υπόψη σε όλα τα ε, επίπεδα της παιδείας και στην ε, επαγγελματική κατάρτιση αλλά και στην εκπαίδευση. Και αυτό να γίνεται συνέχεια, χωρίς διακοπές. Επίσης οι τοπικές και περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και επίσης ε, σε σχέση με τον ε, ε, βιομηχανικό ιστό της οικονομίας θα βοηθήσουν στο να πετύχουμε να γίνει δηλαδή έτσι ένα τρίγωνο μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ τοπικών περιφερειακών αρχών και επίσης Επίσης ε, και με τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ε, αυτά μπορούν να βοηθήσουν την αγορά της εργασίας. Ε, επίσης να υπάρχει ποιότητα, καινοτομία, αποτελεσματικότητα. Είναι κατακλείδη. Η Στατική Ευρώπη 2020 είναι μια πρόκληση, αλλά με την ευκαιρία μπορούμε να βρούμε επαρκείς οικονομικούς πόρους. Να αυξήσουμε το κύρος της ε, κατάρτισης και εκπαίδευσης. Θα προσφύγει ενδιαφέρον επίσης να προβάλλουμε ιστορίες επιτυχίας επαγγελματικής των σπουδαστών και το τι αυξημένο κύρος δίνει σε μια επιχείρηση η σωστή κατάρτιση. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία αναδεικνύω με το κείμενό μου. Όπως προείπα θα πρέπει να είναι σύντομο το κείμενο και να αποφασίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες που αυτές είναι, όσο σας είπα τη γνώμη μου. Στη διάθεσή σας για ό,τι παρατηρήσεις έχετε και για να μου πείτε τις προτάσεις σας για το κείμενο. Hvala za besedo, gospa predsednica. Jaz bom tokrat spet eh, igral vlogo poročevalca v senci in upam, da bom Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά πήρα το ρόλο του σιώδου συζητητή και ελπίζω ότι θα έχω την ευτυχία ξανά να συνεργαστώ με την εισηγήτρια. Ε, χαίρομαι γιατί η Κομισιό προετοίμασε αυτή την ε, νέα πρωτοβουλία, πρωτοβουλία που αφορά την συνεργασία όλων μας για να πετύχουμε τους στρατηγικούς στόχους ενώπιση του 2020. Γιατί θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό. Καταρχάς πιστεύουμε ότι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εργατικού του ιστοδυναμικού ε, που θα έχει πτυχία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίσης, θέλουμε να περιορίσουμε τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Τα περισσότερα αυτά παιδιά προέρχονται από την επαγγελματική κατάρτιση. Γι' αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί η επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα κράτη-μέλη. Ακούσαμε ότι το ποσοστό απασχο... ε, ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο 10%. Επομένως, κάτι δεν πάει καλά με τα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα ποσοστά ανεργίας είναι ακόμα μεγαλύτερα σε ορισμένα επαγγέλματα, για ορισμένα επαγγέλματα. Και από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις χρειάζονται άλλους επαγγελματίες με άλλα προσόντα οι οποίοι όμως δεν υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Άρα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις, στον κόσμο της, ε, να προσφέρουμε στην αγορά ε, κάποια, κάποιους επαγγελματίες, επαγγελματίες τους οποίους χρειάζεται η αγορά αλλά δεν τους έχουμε ακόμα. Οι Υπουργοί Παιδείας θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα στην Μπρούζ και θα προσπαθήσουν να εκπονήσουν μια στρατηγική για τα επόμενα 10 χρόνια. Του χρόνου η Κομισιό και το Συμβούλιο θα ε, εξετάσουν ένα κείμενο το οποίο αφορά και την διαδικασία της Μπολόνια. Επομένως έχουμε δύο παράλληλες αν θέλετε διαδικασίες. Η μία είναι η διαδικασία της Μπολόνια που ε, θα εμπλουτιστεί με νέες απαιτήσει. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια άλλη διαδικασία στον ίδιο περίπου τομέα και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι το 2020 να προχωρήσουμε διότι όπως σας είπα η Ευρώπη θα χρειαστεί εργατικό δυναμικό, θα χρειαστεί άτομα τα οποία να έχουν περάσει από επαγγελματική κατάρτιση. Όμως οι προσπάθειές μας δεν θα στεφθούν με επιτυχία εάν και εφόσον τα κράτη-μέλη δεν συνεργαστούν να εφαρμόσουν κάποια από τα νομοθετικά κείμενα τα οποία έχουν ήδη περάσει και τα, τα οποία έχουμε ήδη ε, αποφασίσει θέματα ε, πρωτοβουλίες για την επαγγελματική κατάρτιση κτλ. Επίσης, εάν δεν εξασφαλίσουμε και χρηματοδότηση κάποιων, κάποιων προγραμμάτων στην επαγγελματική κατάρτιση ε, δεν, θα, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μιλάω για τα προγράμματα όπως το Λεωνάρδο Νταβίντσι, παραδείγματος χάρη. Επομένως, η επαγγελματική κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής για το 2020. Θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν τα σχολεία και θα πρέπει να περιορίσουμε και την ανεργία των νέων. Η ανεργία των νέων αγγίζει το 20% τώρα. Όμως, εάν έχουμε μια αποτελεσματική ή μια αποδοτική επαγγελματική κατάρτιση, το ποσοστό αυτό θα μειωθεί σημαντικά. Επομένως, ε, ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε και με την εισηγήτρια και με εσά, έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Μαρία για την, ε, το σχέδιο νομοδότησης που πραγματεύεται ένα πάρα πολύ σημαντικό και πολύπλοκο θέμα και προσπαθεί να είναι σύντομη Παρά όλα αυτά, ήταν δύσκολο έργο. Την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον στην Γερμανία, το, αυτό που λεγόταν από όλου ήταν ότι η κύριε, ε, εκείνη η κοινωνική ομάδα η οποία κυρίως χάνει ε, από την κρίση είναι οι νέοι. Και πραγματικά είναι... Ε, η, η κατάσταση των νέων και λόγω ανεργίας και λόγω ε, θέσεων απασχόληση οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές η κατάσταση των νέων λοιπόν δεν είναι ικανοποιητική εμείς από σαν Ευρώπη στον τομέα της παιδείας και της διαβίου μάθησης κάτι θα πρέπει να κάνουμε θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ μη, ένα πιο έντομο, έντονο μήνυμα που να λέει ότι Εκείνο που, που λέω ότι πρέπει να προσέξουμε με την έκθεση είναι το εξή. Να μην έχουμε μια έκθεση η οποία λέει ότι στη στρατηγική μέχρι το 2020 θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους και να κάνουμε χίλια δύο πράγματα όταν την σήμερα η μέρα βρίσκονται σε καταστροφική κατάσταση οι νέοι. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια γιατί έδωσε, παρουσίασε ένα πάρα πολύ πλήρες πλαίσιο. Θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα με τους προλαλήσαντες, διότι το μήνυμα πρέπει να δοθεί. Εμείς ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ανεργία για τους ε, νέους που φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 40% και πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξεκινήσουν ε, εκ νέου, αν θέλετε, την ε, επαγγελματική τους καριέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη παίζει το μέλλον της ε, στην, στα, προσόντα, στα επαγγελματικά προσόντα. Επίσης, η Ευρώπη δεν έχει δώσει ένα σωστό παράδειγμα, διότι πολλά προγράμματα κόπηκαν, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες, και αυτό ίσως πρέπει να το πούμε, ότι στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης περικόπτουν ακόμα περισσότερα τα προγράμματα. Αυτό είναι ένα μήνυμα πολύ ισχυρό, το οποίο θα πρέπει να επαναλάβουμε. Επίσης, θεωρώ ότι θα έπρεπε να ξαναμιλήσουμε για τη διαδικασία της Μπολόνια και τη διαδικασία της Κοπενχάγης γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να χαθούν σε σχέση με, την, ε, το θέμα της κινητικότητας και των προσόντων στην Ευρώπη. Ε, πολλά πανεπιστήμια δεν ε, εφαρμόζουν το αμοιβαία αναγνώριση. Επίσης, κάπου σε αυτές τις παραγράφους θα πρέπει να δείξουμε το εξής. Μιλάμε για προσόντα υψηλή εξειδίκευση, προσόντα τα οποία δεν αποκτώνται στο πανεπιστήμιο, και το έχω πει πάρα πολλέ φορές και άλλα μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το θέμα και ίσως στην Γερμανία, στην Αυστρία να υπάρχει μια δομή η οποία να είναι πιο ενοποιημένη τέλος πάντων σε άλλες χώρες σαν τη δική μου χώρα που δεν είναι τόσο καλά οργανωμένα τα πράγματα. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες εκπαιδευτικές αν θέλετε για απόκτηση υψηλών ε, επαγγελματικών ε, προσόντων ανώτερου επίπεδου, αν θέλετε, η συνεργασία ανάμεσα στα ανώτερα ιδρύματα που θα προσφέρουν αυτή την επαγγελματική κατάρτιση και τις επιχειρήσεις. Και εκεί περνάω στην διαβίου εκπαίδευση, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Τελευταία τελευταίο σημείο, τα ευρωπαϊκά προγράμματα Λεωνάρντο πιο συγκεκριμένα, κατά την άποψή μου θα πρέπει να το υποστηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό. Στην ε, στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 λέμε ότι κάθε νέος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ε, εκπαίδευση στην, και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Τώρα όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο, ο Λεωνάρντο και, το, και το πρόγραμμα Έρασμος για τους νέους είναι προγράμματα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να ε, προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Μαρία για την, το σχέδιο έκθεσης το οποίο πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Πέρα από άλλα θέματα που ήδη αναφέρθηκαν νομίζω ότι θα πρέπει κάπου να βάλουμε και το θέμα του δημογραφικού προβλήματος της Ευρώπης βεβαίως υπάρχει οικονομική κρίση και τα λοιπά και αυτό δημιουργεί θέμα απασχόλησης αλλά σε μερικά χρόνια πάρα πολλά άτομα από υψηλά στελέχη και με πολλά προσόντα θα φύγουν από τις επιχειρήσεις, θα συνταξιοδοτηθούν ε, και από, δεν μπορούμε να α, λοιπόν να προχωρούμε χωρίς 40% των νέων όπως ακούσαμε να έχει καμία πρακτική Πήρα δουλειά, διότι είναι άνεργοι. Ή να, να μην προετοιμάζουμε τους ανθρώπους αυτούς για να πάρουν τις θέσεις αυτών που θα συνταξιοδοτηθούν ως Νούπο» είναι ένα σημαντικό θέμα πρέπει να το αναφέρουμε και βεβαίως οι υπουργοί οι οποίοι στην σύνοδό τους ε, έδωσαν κάποια λάθος μηνύματα κάποια άσχημα μηνύματα για το Λεωνάρντο και τέτοιου είδους προγράμματα για μένα αυτό με πονάει ιδιαίτερα πολύ νομίζω ότι ήδη έχουμε κάνει ολόκληρο αγώνα και έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά και να μπορέσουμε να πείσουμε αν θέλετε κάποιους σπουδαστές να πάνε στο εξωτερικό να πάνε να φύγουν από τη χώρα τους ε, είναι δύσκολο και για αυτούς να συνεχίζουν το πρόγραμμα οπότε δεν χρειαζόμαστε τους υπουργού παιδείας να πούν ότι αμφισβητούν ουσιαστικά το μέλλον αυτών των προγραμμάτων. Θα πρέπει λοιπόν και για αυτά τα προγράμματα να πούμε κάτι στην έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Χίρς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης ε, συγγήτρια, αλλά συγγήτρια στην Επιτροπή Απασχόλησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για το σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης, αναφέρθηκαν εδώ ναι, πάρα πολλά πράγματα, ειδικά για την επαγγελματική κατάρτιση, ε, αναφέρθηκε ήδη το πρόβλημα αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Ε, ε, αν ακόμη και αν καταφέρουμε το 15-20% που είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο να το κατεβάσουμε στο 10% κάθε τάξης, κάθε χρονιάς, αυτό θα είναι άθρος. Επίσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν τώρα από το σχολείο αλλά και τα επόμενα 10 χρόνια παραμένουν στη, κατά πάσα πιθανότητα άνεργοι και άρα επηρεάζουν και τα τα, τις μελλοντικές χρονιές αν θέλετε λοιπόν θα πρέπει να δούμε εάν και κάποια σχόλια που έκαναν ε, έκανε για το θέμα αυτό η Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αλλά ένα άλλο ε, ζήτημα το οποίο μου φαίνεται πολύ σημαντικό και δεν συζητήθηκε είναι το image η εικόνα των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτός ο οποίος δεν πάει στο πανεπιστήμιο και ακολουθεί μοναχά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται κάπου από τα μίντια και τα λοιπά υποδέστερος αυτών που ε, αυτού που πάει στην ανώτατη εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε, αν θέλετε, την επαγγελματική κατάρτιση με τα πανεπιστήμια, τόσο ώστε αυτός που έχει κάνει επαγγελματική κατάρτιση κάποια στιγμή να μπορεί να πάει στην ανώτατη εκπαίδευση αύριο. Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό είναι το θέμα των βιογραφικών έτσι ε, και της μονιμότητας σε μια κάποια δουλειά. Άμα δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους από τα βιογραφικά τους, ε, άμα δούμε ε, πως κλείνουν οι επιχειρήσεις πραγματικά δεν μπορούν δεν υπάρχει περίπτωση από εδώ και μπρο κάποιο να πάει σε μια δουλειά στα 30 του και να μείνει εκεί μέχρι να πάρει σύνταξη μιλάμε για πράγματα που είναι πολύ πιο ρευστά, πολύ πιο ελαστικά. Χρειάζεται μια ελαστικότητα και από την πλευρά του εργαζομένου. Χρειάζεται, εδώ εμπλέκονται και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους εργοδότες και από τους εργαζόμενους υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά για να και θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα συνδέσουμε και με το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη φαίνεται να έχει έλλειψη σε ορισμένε ειδικότητε και αυτό είναι πολύ παράξενο. Ε, τώρα για την κινητικότητα είναι παράξενο γιατί ο, πολλοί άνθρωποι δεν φεύγουν από τη χώρα τους γιατί δεν φεύγουν από τη χώρα τους το θέμα της γλώσσας είναι ένα σημαντικό ζήτημα και το άλλο είναι το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων. Με τη διαδικασία της Κοπενχάγης έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με κάποια εργαλεία αναγνώρισης, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνώρισης προσόντων. Παραδείγματος χάρη, το Europass είναι μεγάλη ε, επιτυχία. πολύ... Ε, χρησιμοποιούν τώρα το Europass για να βρουν δουλειά. Αυτό είναι καλό. Και κάτι τι άλλο. Μακάρι να βρίσκαμε ένα άλλο εργαλείο ακόμη για που να περιγράφει τα μαθήματα που ακολούθηκε, ακολούθησε κανείς στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης. Δηλαδή, να, ο εργαζόμενος να ξέρει ότι μπορεί να έχει κάποια προσόντα ε, έχει κάποια προσόντα, έχει μια κάποια δουλειά, να ξέρει ο εργαζόμενος ότι μπορεί να συνεχίσει να μαθαίνει διαβίου να καταγράφονται τα προσόντα του και άρα να μπορεί να ζητήσει και να ψάξει μια καλύτερη δουλειά όταν ξαναμπεί στην ομάδα, στην α, αγορά εργασίας. Η Μαρή Τερέζ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την Μαρία για την ε, έκθεσή της. Νομίζω ότι έχει θίξει τα πιο σημαντικά θέματα κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο στον οποίο ζούμε, πρέπει να προσαρμόζουμε τα νέα μοντέλα, να, προσαρμόζουμε τα παλιά μοντέλα και να δημιουργούμε νέα μοντέλα. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες ε, ε ανάγκες και ικανότητες οι οποίες απαιτούνται. Ε, θα πρέπει όντως ε, να επιστήσουμε την προσοχή, να στράψουμε την προσοχή μας ε, σε κάποια θέματα τα οποία αγνοούμε μέχρι στιγμής, αλλά που στο ευρωπαϊκό χώρο τον οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε θα επιτρέψουν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας. Όταν λέει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την δημιουργικότητα και την καινοτομία θα έλεγα, θα πρέπει στα εκπαιδευτικά μας μοντέλα να σκεφτούμε και αυτόν τον τομέα καινοτομία, διότι μέχρι στιγμή έχουμε παραμείνει σε κλασικά πρότυπα και από αυτά θα πρέπει να ξεφύγουμε. Επίση, η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση θα πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο, θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερο γόητρο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γόητρο και το λέει και η συγκήτρια στην έκθεσή τη. και δημιουργία γεφυρών ανάμεσα στην, ε, στις επιχειρήσεις ε, και στο, στην ανώτατη εκπαίδευση, διότι δεν θέλουμε βέβαια και η ανώτατη εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση να, να προσανατολιστεί αποκλειστικά και μόνο στην, ε, στις επιχειρήσεις, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και επίσης υπάρχουν και αυτές οι εγκάρσιες στρατηγικές ή πολιτικές Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, πάρα πολλά σχέδια τα οποία προτείνει η Ευρώπη και όχι μόνο στον τομέα της εκπαίδευση και της κατάρτισης μπορούν να βοηθήσουν. Ευχαριστώ. Να κάνω κι εγώ δύο παρατηρήσει, λέει πρόεδρος. Πρώτα πρώτα να επιθυμίσω ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι θετό παιδί αν θέλετε της παραδοσιακής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάποιο, η Μαρία λέει ότι πραγματικά καλό θα ήταν να βάλουμε εδώ παραδείγματα και ε, ιστορίες επιτυχίας για την επαγγελματική κατάρτιση. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις χώρες που υπάρχει μαθητεία, που ανέκαθεν υπήρχε ε, ε, έντα, δινόταν προσοχή στην επαγγελματική κατάρτιση, η ανεργία είναι χαμηλότερη στη Γερμανία, στην Αυστρία. Η, η υπάρχουν ε, εναλλακτικέ λύσεις με την επαγγελματική κατάρτιση και τη μαθητιακή οι νέοι έχουν ακριβώς αυτές τις, επιλογές και γι' αυτό δεν έχει ε, έχουν περισσότερες επιλογές. Χρειαζόμαστε με 40, μας λείπουν 40% ή χρειαζόμαστε 40% ειδικευμένους εργαζόμενους, ή εργάτες. Δεν λέει πουθενά ότι αυτοί πρέπει να, να έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν τελειώσει ένα τεχνικό λύκειο οι άνθρωποι αυτοί, να έχουν κάνει μια επαγγελματική κατάρτιση. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θα πρέπει να προσέξουμε τέτοιου είδους καλές πρακτικές που ισχύουν σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, να τις προωθήσουμε και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό το σημείο 8 της έκθεσης της Μαρίας θα πρέπει να το εμπλουτίσουμε. Μετά, αναγνώριση, αμοιβαία αναγνώριση κάποιων επαγγελμάτων. Στο Λουξεμβούργο να σας πω, στη γειτονική μου χώρα, γιατί εγώ είμαι στο ΣΑΡ, στη Γερμανία δίπλα μας είναι, λοιπόν στο ο, ορισμένα επαγγέλματα όπως παραδείγματο χάρη η φροντίδα των ηλικιωμένων δεν αναγνωρίζεται ως επάγγελμα. Στη Γερμανία υπάρχει το επάγγελμα αυτό ε, και έχουμε φροντίδα των ηλικιμένων υψηλού επίπεδου, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που υπάρχει μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων που έχουν διάφορες μορφές άνοιας. Οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν και στο Λουξεμβούργο. Μπορεί να πάνε και οι Γερμανοί να δουλέψουν στο Λουξεμβούργο σε αυτή την ειδικότητα, αλλά πληρώνονται λιγότερο, διότι δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμά τους. Δεν είναι δυνατόν το πρόβλημα αυτό να είναι Λουξεμβούργοι Ιταλιανό, γερμανικό πρόβλημα μονάχα. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό. Και τέτοιου είδους προβλήματα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το βάλει στην εκθεσή της η Μαρία αυτό, αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Και μια ερώτηση Μαρία, στο σημείο 5, προώθηση της δημιουργικότητας. Τι θα πει αυτό, ενίσχυση της ε, δημιουργικότητας στο σημείο 5 δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ε, ε, αν εννοείς ε, να μπορεί κα... η δημιουργικότητα τουλάχιστον στα γερμανικά δεν λέει τίποτε. Θα έπρεπε να λέμε ίσως αυτονομία εδώ και ανάληψη πρωτοβουλίας. Αυτό ναι. Η Κομισιόν θέλει κάτι να πει, κύριε Ρεγκάλντο. Κύριε Ρογκάλντο δεν είναι εδώ. Ναι. Äh, Ο κύριο Δελκάδο, όχι. Ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα μοναχά να πω ότι είμαι σκιώδη για την Επιτροπή ανάπτυξη για, για το θέμα αυτό και θα ήθελα να κάνω μια-δυο παρατηρήσει. Η ο κλάδος δημιουργικών επαγγελμάτων, creative ε, στην Ευρώπη είναι αρκετά προωθημένος το Riverdance θα ξέρετε γιατί μιλάω ήταν μεγάλη επιτυχία και δείχνει τη δυνατότητα να πάρει κανείς ένα πολιτιστικό προϊόν και να το αναπτύξει και να το προωθήσει για το 6-6 μιλάς. Είμαστε ακόμα για το 6 μιλάς. Της ημερήσιας διάταξη μιλάς. Είμαστε στο 5 λέει η πρόεδρος. Sorry λέει ο κύριος Κέλλη. Commission please. Thank you, Chair. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαιρόμαστε που ακούσαμε όλα τα σχόλια αυτά σήμερα αλλά ε, και ευχαριστούμε και για το σχέδιο της έκθεσης και εμείς τα ίδια πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την κρίση που ζούμε και στην ε, ανεργία αυτή η έλλειψη αντιστοιχίας ανάμεσα στα στις επαγγελματικές ανάγκες και στην εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θίξατε, Πρόεδρε, και το πρόγραμμα της Γερμανίας, που είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα, αλλά και η διαβίου επαγγελματική κατάρτιση ε, και με την ε, αύξηση ηλικία του, του πληθυσμού υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Το πρόβλημα της διαπερατότητας ε, είναι πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα είναι, μάλλον το καλύτερο σύστημα για την επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτό το οποίο επιτρέπει να γίνονται ανταλλαγές ανάμεσα σε διάφορα συστήματα εκπαίδευσης και, στην, στον επαγγελματικό κόσμο. Εάν θέλουμε οι νέοι να πάνε σε επαγγελματική κατάρτιση, θα πρέπει να τους ε, δείξουμε ότι μπορούν από εκεί να πάνε και στο πανεπιστήμιο αν θέλουν. Γιατί αλλιώς δεν θα ε, επιλέξουν επαγγελματική κατάρτιση. Συμφωνώ απόλυτα ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα τρόπο για να περιορίσουμε τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν τα σχολεία, όμω πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου, υψηλή ποιότητα. Ε, εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα είναι εναλλακτική λύση για τα παιδιά αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν ε, οι υπουργοί στην Μπρούζ. Το μήνυμα σας υπάρχει και του χρόνου θα πρέπει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να, να εργαστούν για να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις αρχές που θα αποφασίσουν οι Υπουργοί και εκεί θα χρειαστώ τη συνεργασία σας, διότι θα πρέπει και η Γερμανική κατάρτιση να ε, συνδεθεί και με τους άλλους τομείς της παιδείας. Και το σημερινό, νομίζω, παράδειγμα είναι να ε, μας δείχνει ακριβώς πώς μπορούμε να δουλέψουμε και στο μέλλον. Πρόεδρος, ένα λεπτό. Θα ήθελα να απαντήσω το εξή. Δεν πιστεύουμε ότι αυτά τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο και που θέλουμε να μειωθούν ως προς τον αριθμό τους θα τελειώσουν κάποια στιγμή το σχολείο και μετά θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Δεν, κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούν. Αυτοί, αυτά τα παιδιά χρειάζονται μια επαγγελματική κατάρτιση. Δεν είναι ντροπή να πούμε ότι το ΒΕΤ που είναι μία πόρτα, μία ε, πύλη προς την ανώτατη εκπαίδευση αλλά η χρησιμοποίηση του συστήματος ΒΕΤ δεν είναι ε, του ΕΕ κάπα που λέμε στα ελληνικά επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση η χρησιμοποίηση αυτού αυτών των εργαλείων ε, δεν είναι η λύση την οποία προκρίνουμε για τα παιδιά αυτά. Η συγγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι για τη συζήτηση που έγινε. Γιατί βλέπω ότι τα μέλη της ε, Επιτροπής ε, συμμερίζονται τις ε, απόψεις μου, αλλά και την ανησυχία μου για τους νέους. Διότι οι νέοι είναι που πλήττονται από, τον, ε, από την ανεργία. Εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε μια γενιά στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Και για τους νέους, αλλά και για, τους, και για την Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, τις, ε, για τη συνεισφορά σας. Ήταν πολύ χρήσιμες όλες τις παρατηρήσεις που άκουσα. Όταν ε, αποφασίζουμε κάποιους κανόνες, προφανώς ε, θα υπάρχουν κενά. Η έκθεση πρέπει να είναι περιορισμένη. Έχουμε και ένα περιορισμό στον αριθμό των χαρακτήρων που θα πρέπει να έχει μια έκθεση. Αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όλα τα σχόλια. Όμως αυτό το οποίο υπάρχει στην αρχική έκθεση δεν πρέπει να το επαναλάβουμε. Γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε μια ποιοτική έκθεση στο τέλος της ημέρας. Όταν μιλάμε για δημιουργικότητα, ε, θέλουμε να, έχει κάποιο, να έχουμε την ικανότητα να αποφασίσουμε να επιλέξουμε την καινοτομία. Αυτό ίσως να μην συμβαίνει σε όλες τις χώρες, ε, αλλά σε κάποιες χώρες ε, η εκπαίδευση ήταν ιδιαίτερα παθητική. Διδάσκαμε, διδάσκουμε κάποια πράγματα στον κόσμο, όμως δεν, τους, μαθαίνουμε στα παιδιά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Άρα δεν θα πρέπει τα άτομα να είναι παθητικά, το ανάποδο, πρέπει να γίνουν δραστήρια. Δηλαδή, εγκαταλείποντας την επαγγελματική κατάρτιση, το πανεπιστήμιο, τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να στηρίζονται στις ιδέες τους. Δεν ξέρω τώρα αν η δημιουργικότητα είναι η σωστή λέξη θα μπορούσαμε αντί για δημιουργικότητα να πούμε ότι συστήνει, συνιστά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης περιλαμβανομένης και της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης την ενίσχυση της πλήρους α, εκμετάλλευση των ικανοτήτων τους ή του δυναμικού τους να να μπορεί το παιδί, ο νέος, να ακολουθήσει και ε, ε, δρόμους και πορείες που δεν είναι παραδοσιακοί. Τι να σας πω, να πάει να στήσει μια μικρή επιχείρηση. Λοιπόν, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου μοναχά, την επόμενη Τρίτη δηλαδή. Γιατί θέλουμε να τελειώσουμε, να είμαστε έτοιμοι ε, και να ψηφίσουμε το Γενάρη. Η Επιτροπή Επασχόλη θα ψηφίσει το Μάρτι. Α, για να ψηφίσουμε όμως το Γενάρη πρέπει να υποβάλουμε τροπολογίες μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Προχωρούμε στο σημείο 6 της σας διάταξης. Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Τώρα είναι το θέμα αυτό. Μαχίτε Χάισε Σάντσες Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου επιτρέψετε να ε, συζητήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και τον Γενάρη. Η Κομισιόν δημοσίευσε πριν από μερικούς μήνες μία πράσινη βίβλο σε αυτές τις, ε, σε αυτές τις βιομηχανίες δημιουργικές και πολιτιστικές που και εκεί δημιουργήθηκε μία συζήτηση για το πώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι βιομηχανίες οι δημιουργικές και οι πολιτιστικές. θα πρέπει να βρούμε μέτρα ε, και πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν, ε, θα επιτρέψει αυτός ο κλάδος να ε, προχωρήσει, να προωθήσει, λαμβάνοντας υπόψη και τις, την περίοδο την οποία διανύουμε. Αυτή, αυτός ο κλάδος παρουσιάζει μια καινοτομία, παρουσιάζει δυνατότητες δημιουργίας θέσης απασχόλησης, προσφέρει δυνατότητες μιας βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομίας. θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, πιστεύω, για το κατά πόσο θα πρέπει να βρούμε έναν ορισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων που καλύπτουν αυτούς τους όρους κλάδος του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Θα ήθελα να υποστηρίξω και να τονίσω το γεγονός ότι αυτές, αυτός, αυτός ο κλάδος ε, έχει ένα ε, ε, δυναμικό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα. Το 2,6% του ΑΕΠ καλύπτει αυτός ο κλάδος και προσφέρει απασχόληση σε περίπου 5 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη των 27. Πέραν της άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ, ο κλάδος αυτός είναι ένας κινητήρας καινοτομία και κοινωνικής πρόοδου σε πάρα πολλούς τομείς. Για να μπορέσει αυτός ο κλάδος, ε, αυτή η κλαδή τέλος πάντων, να εποφεληθούν καλύτερα από την πολιτισμική ποικιλομορφία, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση που είναι ο κινητήρας ε, της ανάπτυξης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα μέτρα μέσα και να βοηθήσουμε αυτό το κλάδο να προχωρήσει στο τοπικό και περιφερειακό πλαίσιο, διότι ο πολιτισμός είναι και ένα μέσον περιφερειακής ανάπτυξης. Το θίξαμε αυτό το θέμα και για την εκπαίδευση. Μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες, ε, σε, ε, στην ανάπτυξη μιας περιοχής και, στην, ε, και στο χώρο της μιας περιοχής. Όλα αυτά τα στοιχεία, έστω και αν είναι ανεπαρκή, θεωρώ ότι είναι αρκετά για να προσανατολίσουμε κάπως τη συζήτηση και να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας, έτσι ώστε οι πολίτες μας να έχουν μια πιο εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό σε διάφορους κλάδους που τους στους οποίους απασχολούνται. Θα πρέπει να καταρτήσουμε μια στρατηγική έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και μια κοινωνική συνοχή σε αυτή την προοπτική η πράσινη βίβλος αναφέρει πολλές ε, δυνατότητες. Ε, δυνατότητα πειρασματισμού και καινοτομίας, ε, προσόντα, πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ο συνδυασμός όλων αυτών μπορεί να αυξήσει το πολιτιστικό και οικονομικό δυναμικό μιας περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια ευκαιρία για τους καλλιτέχνες μας να λάμψουν στο... σε διεθνές επίπεδο. Και βέβαια σε όλους τους τομείς ε, μιλάμε και για τη χρηματοδότηση, διότι η χρηματοδότηση είναι κάτι σημαντικό και εξαρτάται από την καλή χρήση των ε, μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, θα πρέπει να γίνει μια σωστή διαπραγμάτευση ανάμεσα στους ιδιωτικούς και δημόσιου φορείς και σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουμε να προασπίσουμε την ε, ε, πολιτισμική διαφοροποίηση. Τώρα, η ψηφιοποίηση. Ε, βλέπουμε ότι εδώ χρειάζεται μια συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Το πνεύμα των, της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι μια συνεργασία δυναμική Μιλάμε και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης που μπορούν να προσφέρουν στον τομέα όλη την, ε, όλο το δυναμικό καινοτομία τους. Επομένως θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις, αυτόν τον κλάδο και να ε, επιβάλλουμε την δίκαια αμοιβή της ε, δημιουργίας, της πολιτιστικής δημιουργίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θα πρέπει να, να προστατεύσουμε τους καλλιτέχνες μας από την πειρατεία εδώ και δέκα χρόνια μιλάμε πολλές φορές ε, για την ε, οικονομία του άειλου, για την κοινωνία της γνώσης, για την ε, σημασία που έχει η στρατηγική της Λισαβόνας, για μια ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης. Αυτές οι συζητήσεις έγιναν σε διάφορους κύκλους πολιτικούς, σε ακαδημαϊκούς, στην κοινωνία των πολιτών, για να βρούμε νέες μορφές οικονομίες, για να βρούμε νέους, νέες μορφές ρύθμισης θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσεις. Από όλη αυτή τη συζήτηση ήθελα να πω ότι ε, το γόητρο και η έλξη του δωρεάν ε, δεν ε, Δεν, δεν, δεν υπάρχει πλέον, κυρίως όσον αφορά το πολιτιστικό προϊόν και για την δημιουργία του και για την κατανάλωσή του. Οπότε είναι αλήθεια ότι άλλαξε ε, άλλαξαν τα πράγματα και το θέμα της αμοιβή των δημιουργών και η αξία του περιεχομένου είναι τώρα στο επίκεντρο των πραγμάτων και αυτό το, το χαιρετίζουμε και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι η ψηφιακή δημιουργία νόμιμη και πώς θα ε, ωφεληθεί ο πολιτικός τομέας από πλευράς οικονομικής και για αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική και την πολιτιστική, να εκπαιδεύσουμε το κοινό του της, της αύριο και επίσης αυτή η νέα οικονομία να γίνει σεβαστή και όλοι είμαστε βυθισμένοι σε οικονομική κρίση και έχουμε επομένω κάποιες πρωτοβουλίε ώστε να, να τονώσουμε κάποιου τομείς για τη ζωτικότητά τους ε, είναι αξιοθαύμαστε και επίσης θα πρέπει η Επιτροπή να προβληματιστεί και συμφωνώ με τη γενική διαπίστευση ότι η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση είναι σημαντικές για την δημιουργία, όμως η ανάλυση της πράσινης βίβλου δεν είναι υπαρκής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κινητοποιηθεί για να προστατεύσει την καλλιτεχνική δημιουργία και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η πολιτικός τομέας θα, θα πρέπει να ε, προσεχθεί, να αναβαθμιστεί και να προσαρμοστεί στην ψηφιακή τεχνολογία. Το, το, θα πρέπει η αγορά να είναι επικερδής. Θα πρέπει να υπάρχει πραγματική και πολύμορφη προσφορά καλλιτεχνική. Συνεχίζει και διαβάζει ο μιλήτρια γρήγορα. Οπότε θα πρέπει επομένω να επιμείνουμε όσον αφορά την σχέση μεταξύ ε, πολιτιστικής δημιουργίας ε, και... για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς δουλεύουν αυτές οι τρεις μεταβλητές και για αν βοηθούν ή δεν βοηθούν την δημιουργία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σταθούμε στον ρόλο τους ως φορείς ε, της οικονομίας ε, και καλά τα λέει εδώ η πράσινη βίβλος. Όμως θα έπρεπε να προβληματιστούμε όσον αφορά τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να έχουμε μαζική προσφορά υπηρεσιών περιεχομένου πολιτιστικού online και στα πλαίσια αυτά ζητώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβληματιστεί όσον αφορά το συντελεστή ΦΠΑ για τις πολιτιστικές online υπηρεσίες. Πλουραλισμός στην ε, διάδοση της μουσικής ή του, του, βίντεο και έτσι να έχουμε ε, την αναζήτηση ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικού όσον αφορά την, την online ε, διάχυση αυτών των έργων και να είναι και το φορολογικό περιβάλλον ευμενές. Είναι διτή η υφή αυτών των έργων, ε, θα υπάρχει κοινωνική αξία και συμβολική και δεν θα πρέπει μόνο να διέπεται η πολιτιστική αγορά από, από τους κανόνες της αγοράς και αυτό φάνηκε και από την κρίση ε, ενώπιον της οποίας η δημιουργία, η, ο πολιτισμός, ε, έχει δείξει ότι έχει στέρεες βάσεις με τις εκδηλώσεις του, όμως θα πρέπει να κάνουμε βήμα παραπάνω και να προσαρμόσουμε το ρυθμιστικό περιβάλλον και έτσι να έχουμε μια πλατφόρμα προβληματισμού, ανταλλαγή αρίστων πρακτικών ούτω ώστε να δούμε πώς θα έχουμε πολιτιστική παγκοσμιοποίηση στα πλαίσια της ε, σύμβασης της ε, UNESCO. Είναι το πιο σωστό το πώς έτσι θα αξιοποιήσουμε την πολιτική κληρονομιά. Να μην μας νοιάζει μόνο το, το, το αύριο, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι να πηγαίνουμε πιο πέρα στο μέλλον. Ευχαριστούμε Μαρή Τερέζα, αλλά όταν κανένα διαβάζει είναι δύσκολο και όταν διαβάζει δύσκολο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και ευχαριστούμε τους ναι, Ναι, με συμπαθάτε με λέει η Μαρή Τερέζ. Formidable. Bon. Ah, αλλά, αγαπητή Μαρή Τερέζ, εντάξει αυτό τώρα, αλλά Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια πράσινη βίβλο για τα θέματα αυτά αυτό είναι καλό και ζήτησε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν την πράσινη βίβλο και να απαντήσουν. Αυτό που κάνουμε λοιπόν εδώ τώρα είναι να απαντήσουμε ακριβώς την πράσινη βίβλο της Κομισιόν. Α, αν έχουμε καινούργιε ιδέες που δεν τις έχει βάλει στην πράσινη βίβλο της Κομισιόν, να τις πούμε τις ιδέες. Αν έχεις το πρόβλημα με το ΦΠΑ, βεβαίω να το πούμε και να δούμε αν μπορεί να περάσει ή όχι. Ποιος θέλει τώρα το λόγο, η κυρία το λογο Κώστα. Ringrazio comunque E Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρή Τερές και για το πάθος της αλλά και για την δουλειά που έκανε. Είναι χρήσιμο να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτή την πράσινη βίβλο, διότι αποτελεί μια πρόκληση, όχι μονάχα για την ε, δικιά μας Επιτροπή, αλλά και για όλο το Κοινοβούλιο. Διότι θεωρώ ότι η πράσινη βίβλος αποτελεί μια ευκαιρία να αναρωτηθούμε αυτός ο κλάδος του πολιτισμού και της δημιουργιότητας στην Ευρώπη ποιο είναι. Διότι αυτός ο κλάδος έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Γιατί ε, από αυτόν εξαρτάται πώς βλέπει ο κόσμος στην Ευρώπη, από το πολιτιστικό προϊόν και από την δυνατότητα καινοτομία που έχει. Και αυτό θα πρέπει να, αυτή είναι μια πτυχή που είναι πάρα πολύ σημαντική και για την στρατηγική του, της Ευρώπης το 2020. Δηλαδή θα πρέπει αυτή αυτό το σημείο να ενταχθεί στην στρατηγική της Ευρώπης 2020, ε, 2020. Η Κομισιό το απαντώντας σε 300 κάτι ερωτήσεις, ε, το, ε, το εξακρίβωσε και στη χώρα μου, δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, κάποιες ερωτήσεις. Μήπως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι ο πολιτισμός είναι ένα κοινό αγαθό. Επομένως, το οποίο ανήκει σε όλους εννοώ. Επομένως, μήπως θα πρέπει και οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν περισσότερο για να προωθήσουν ε, τον πολιτισμό, αλλά και αγαθά τα οποία αποτελούν ε, μέχρι στιγμής ε, παρέμβαση, αντικείμενα παρέμβασης μόνο του δημόσιου τομέα, αλλά θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη. Θεωρώ ότι το πράσι, η πράσινη βίβλος αναφέρει 8 τομείς, πάρα πολύ σημαντική. Πολλές παρατηρήσεις που, μου, που έχω δει εγώ ε, είναι περιοριστικής. Ας πούμε ένας τομέας όπως η μόδα, και ο πολιτιστικός τομέας επίσης, ο τουρισμός επίσης ε, που αποτελεί τη σύνθεση πολλών ε, στοιχείων ε, καινοτομία και που παρουσιάζει μεγάλη, μεγάλες δυναμικότητες διότι αντιπροσωπεύει την, τον πλούτο αν θέλετε του, της υπήρου μας. Αυτά μήπως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε. Δεύτερον, η, η, εξειδίκευση αν θέλετε αυτού του κλάδου σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Το αναφέρει, αλλά πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Η πολιτιστική, ο κλάδο αυτό τέλο πάντων του πολιτισμού μπορεί να ενταχθεί όχι μονάχα εδώ, με στα πλαίσια αυτής τη ενέργεια, αυτή τη δράση, αλλά θα μπορούσε να ενταχθεί και σε άλλα προγράμματα. Π.χ. το πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την έρευνα και τη βιομηχανία. Μιλάω για τα ταμεία, τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρώπης Θα πρέπει να εντοπίσουμε συσχετισμούς και δυνατότητες σύνδεσης και με άλλα προγράμματα. Αυτή η αλληλεπίδραση και αυτή η σχέση θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο. Και τρίτον, το θέμα της κινητικότητας των ε, καλλιτεχνών, των έργων ε, κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι εγκάρσιο επίσης και αφορά δηλαδή και άλλα προγράμματα αυτή, αυτός ο εγκάρσιος χαρακτήρας, ο οριζόντιος χαρακτήρας θα πρέπει να τονιστεί και θα πρέπει να τονιστεί και η ιδιαιτερότητα του κλάδου. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι, οι, επιχειρήσεις που ε, δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα είναι πάρα πολύ μικρές. Μιλάμε για μικρά γραφεία, για στούντιο αν θέλετε, που, ε, για, ε, γραφεία μελετητικά κτλ. που απασχολούν πολύ λίγα άτομα και μιλάμε και για συγκεκριμένες ε, ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Άλλα πράγματα ο οπτικοακουστικός τομέας, άλλος ας πούμε ε, ένας άλλος δημιουργικός τομέας. Ε, μια άλλη ιδιαιτερότητα που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι ότι έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του καθεστώτος που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μικρές. Επίσης, το θέμα του καλλιτέχνη, του δημιουργού. Το έχουμε δει πολλές φορές συζητώντας εδώ με συγγραφείς, με καλλιτέχνες, με, με δημιουργούς γενικότερα. Θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάρτιση, η εκπαίδευση των ατόμων δεν είναι η επίσημη, δεν είναι η τυπική, είναι άτυπη πολλές φορές. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ένα ερώτημα που αφορά όλο τον κλάδο αυτόν. Η πρόκληση της ψηφιοποίησης αυτό σημαίνει ότι θα προβλέψουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποια μέτρα τα οποία σήμερα δεν εγκρίνονται σε κάποια κράτη-μέλη διότι θεωρούνται ότι είναι κρατικές επιχορηγήσεις. Ας πούμε, προσφέρουμε δυνατότητες πρόσβασης και διανομής με χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο όπως επίσης και προώθηση στο εξωτερικό όλων, όλης της παραγωγής μας. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον παραγωγή και όχι σαν κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μεγάλο αίτημα από πλευράς άλλων χωρών, ακόμα και της Κίνας, να γνωρίσουν λίγο παραπάνω ε, μαθήματα design, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε να το προωθήσουμε αυτό. Συνολικά όμω, όχι κατακαιρματισμένα. Διότι νομίζω ότι υπάρχει ζήτηση, άρα θα μπορούσαμε να συντονίσουμε και την προσφορά. Vielen Dank. Äh, Herr Kelly, jetzt, jetzt können Sie. Τώρα έχετε το λόγο κύριε Κέλλη. Uh, Συμπαθάτε με. Για πριν αλλά έπρεπε να κουβεντιάσω κάτι με τον συνεργάτη μου και ήμουν αφηρημένο. Σας ευχαριστώ πάντως. Τα περισσότερα τα καλύψατε, να μην λέω τα ίδια. Αλλά ξέρετε, είμαι σκιώδη εισηγητή σε άλλη επιτροπή και διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητε μας για τις αντισώμενες ε, βιομηχανίε και όπως είπαμε και προηγουμένως έχουμε το Riverdance, αυτό το οποίο βγήκε από ένα δίλεπτο νούμερο πριν από 20 χρόνια στη Eurovision και εξελίχθηκε σε πολιτιστική βιομηχανία παγκόσμιου βεληνικού. Να, τι ικανότητε μπορούν να υπάρχουν, τι δυνατότητες υπάρχουν. Και πάρα πολύ. Όταν μιλούν για κουλτούρα και πολιτισμό θεωρούν ότι είναι κάτι κρατικοδίαιτο που πληγωδείται από κράτο και όκ είναι έτσι, είναι βιομηχανία απτυσσόμενη. Επίσης, τα φεστιβάλ. Οι φορές δυνατότητε μπορούν να βοηθήσουν και σε τουρισμό, ε, να διαδώσουν την κουλτούρα, ακόμα και σε μη προνομίχε περιοχές, μειονεκτούσε, παντού στην Ευρώπη. Και αυτό σημαντικό. Ε, και οι καστικές τέχνες επίσης νομίζω ότι εύστοχα αυτά τα έθιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέρσι στο Μανχάιμ είχαμε πάει με την Περιφερειακή Επιτροπή για κάποια μέρη του στόχου 2 και κάπου πήγαμε σε ένα κτίριο για μουσικές δραστηριότητε, νέοι, συγκροτήματα, διαφορετικά είδη μουσικής, διαφορετική προέλευση συνέθεταν μουσική, του παρουσιάζουν και επίσης ακόμα και μουσικό όργανα κατασκεύαζαν. Να, άλλη μια ιδέα. Όλα αυτά δείχνουν πόσο μπορούν να γίνουν στα πλαίσια του πολιτισμού καινούργιες βιομηχανίες. Και φυσικά όλα αυτά βοηθάνε στην πολιτιστική πολυμορφία στα πλαίσια της του 2020 βοηθάτε από όλα αυτά η οικονομία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μπίσκι. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο έχω μια παράκληση. Η έκφραση κλάδι πολιτισμού και δημιουργικότητας, όρος αυτός παραπλανεί. Η πολιτική που ασχολούνται, αυτοί που ασχολούνται με τον πολιτισμό θα πρέπει δηλαδή να πέσουν στα γόνατα και να θαυμάσουν τους δημιουργούς. Λάθος διότι υπάρχουν και πολιτιστικά αγαθά τα οποία είναι πρωτόγωνα ή έχουμε συγκαστικές τέχνες τους πριμιτίφ, τους ναΐφ, να σας την ζωγραφική πόσα λίγα από τα γερμανικά ταλέντα στη ζωγραφική μπορούν και ζουν από την τέχνη τους είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι ζωγραφίζουν μεν και μάλιστα πάρα πολύ ωραία, αλλά έχουν και μια άλλη δουλειά για να επιβιώσουν. Υπάρχουν όμως και και άλλη, υπάρχει βέβαια και μια άλλη πτυχή η οποία δεν είναι καθόλου ε, δημιουργική ε, αυτός ο οποίος ε, για να κάνει λεφτά βάφει σαν να έβαφε και όχι να ζωγράφιζε. Είναι αυτό δημιουργικό στη μουσική. Υπάρχουν, γίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι δημιουργικά όλα αυτά που βλέπω στις διάφορες οθόνες τολμώ να προτείνω πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ δημιουργικά μπορεί να ε, ε, τέλος πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά που γίνονται σε αυτούς τους κλάδους που περιγράφηκαν εδώ να τα θεωρήσουμε δημιουργικά. Άρα ο όρος αυτός ο οποίος δημιουργεί, ε, ο οποίος φαίνεται να έχει εμπεδοθεί στην Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι είναι και αυτό μια πρόκληση ε, να αλλάξουμε τον όρο για την περιγραφή των κλάδων αυτών. Ο σοβαρός τύπος όλο και περισσότερο ε, χρησιμοποιεί τον όρο αυτό βεβαίως ε, μέχρι τώρα θεωρούν του και δημοσιογράφοι δημιουργοί και ο φωτογράφος για, το, για τις ε, εφημερίδες, επίσης καλλιτέχνες. Ε, δεν νομίζω ότι ε, ισχύει αυτό και οι περισσότερες εφημερίδες ε, βλέπουμε ότι ε, όλο και περισσότερο δεν χρησιμοποιούν τον όρο στην προκήρυξη θέσεων παραδείγματο χάνει και τα λοιπά. Ας δούμε λιγάκι πιο ρεαλιστικά το θέμα. Ε, εγώ λέω να βοηθήσουμε τους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας, αλλά να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εισηγήτριά μας έθεσε ένα ευρύ πλαίσιο για να παρουσιάσει το επιχείρημα, το θέμα, γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες παρέμβασης και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον όλων για αυτό το θέμα, όπως το ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε αφορά τις πρώτες σελίδες της πράσινης βίβλου της Κομισιό. Η Κομισιό λέει εκεί ότι εφόσον αυτός ο κλάδος του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ε, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί περισσότερο τις δυνατότητε του, θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή του. Και ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Θα πρέπει να βοηθήσουμε στον κλάδο αυτό να αναπτυχθεί σε τοπικό και σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιβάλλει την παρουσία και τη δύναμή του. Τώρα πώς θα γίνει όμως αυτό? Κάποια θέματα, κάποια πράγματα ακούστηκαν ήδη από τους προαλήσαντες συναδέλφους, δεν θα τα επαναλάβω. Όμως, μια και πρόκειται για πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε και για να επιστρέψω σε μια συζήτηση που κάναμε και πριν από λίγα λεπτά, στο θέμα της κατάρτισης. Διότι πρόκειται για κλάδος που έχουν ανάγκη την εκπαίδευση και την κατάρτιση για να μπορέσουν να προσελκύσουν κάποια άτομα, κάποιους δημιουργούς. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την μεταβίβαση της γνώσης. Γιατί πολλές φορές η γνώση αυτή είναι, αν θέλετε, σε βιοτεχνικό επίπεδο. Είναι μια γνώση, μια, ε, ε, είναι μια πληροφορία η οποία περνάει από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό το λόγο, ταυτόχρονα θα πρέπει να προωθήσουμε όλο το θέμα των, της ανταλλαγής και της δυνατότητας πρακτικών γνώσεων. Πρόγραμμα έρασμος για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Όπως και η δυνατότητα να εποφεληθούμε, να εκμεταλλευτούμε από όλες τις ανταλλαγές των νέων, τα προγράμματα ανταλλαγών νέων, που μπορούν να επωφεληθούν από το έργο αυτών των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου. Δεν θα πω περισσότερα πολλά παραπάνω, διότι ούτω ή άλλως έχουμε την δυνατότητα να τα ξανασυζητήσουμε τα θέματα όταν υποβάλουμε τροπολογίες, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να προσέξουμε και την ε, κατάρτιση και την ε, μεταβίβαση ε, της γνώσης, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να παραμείνουμε σε θεωρητικό επίπεδο αφενός ή αφετέρου να μπούμε σε πολύ συγκεκριμένα θέματα χωρίς να δούμε το γενικό πλαίσιο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κραμπ από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσω σε σχέση με το πώς βαδίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να αναλύσουμε επί τη βάση των αντιδράσεων στο, στο, στο, στο βιβλίο. 350 ήταν οι απαντήσει απαντήσεις ε, στην Πράσινη και, και μέσω του website οι περισσότεροι ήταν ε, διάφοροι φορείς, περιφερειακοί, εθνικοί κλπ. Και επίσης διάφοροι δημόσιοι φορείς Πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν το ότι είχαμε μεγάλη ποικιλία ανά κλάδο, όπως και ανέφεραν οι απόψινοί αγορητές, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, από παντού υπήρξε ενδιαφέρον. Πολύ πάρα πολύ αυτή η κατανομή. Οι περισσότεροι δε, από αυτοί που απάντησαν, είναι από τέχνες και ε, από του χώρους θεάτρου, χορού και λοιπά και επίσης από τα μίδια. Τον Ιανουάριο ξεκινάμε την επεξεργασία του εγγράφου εργασία την ανάλυση επιβέστων των απαντήσεων που έχουμε λάβει και ο στόχο είναι κατά τα μέσα τη επόμενη χρονιά να προχωρήσουμε στην έκδοση ανακοίνωση όπου θα έχουμε προτάσεις πιο συγκεκριμένες για την πολιτική που θα χαράξουμε, για το πώς θα έχουμε ένα πάρα πολύ θετικό περιβάλλον για τις δραστηριότητε αυτές. Σε αυτή τη φάση δεν ωφελεί να μιλήσω για τις λεπτομέρειες των απαντήσεων, αλλά κάτι που θα σας ενδιαφέρει είναι να σας πω ότι πάρα πολλοί μας απάντησαν, είπαν ότι ο κάθε καλλιτέχνης, ακόμα και για έναν τομέα που φαίνεται ότι είναι πολύ εμπορευματοποιημένο είναι η δημιουργία, το ταλέντο, οι δημιουργικοί άνθρωποι. Αυτό το είπαν πολλοί από αυτούς που απήντησαν. Ήταν ο κοινός προνομαστής όλων αυτών. Το άτομο, το, το πρόσωπο, το δημιουργικό. Και δεν θέλουμε εδώ να έχουμε κάποιο τεχνητή, τεχνητή διάκριση μεταξύ αυτών και των πετυχημένων εμπορικών δραστηριοτήτων, γιατί το ένα είναι προπόθεση του άλλου, άρα θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη έχει χαράσει μια πολιτική. Αλλά όπω είπαμε, για το πρώτο ήμιση του Ιανουαρίου θα δημοσιοποιήσουμε αυτό το έγγραφο, θα αναλύσουμε όλε τι απαντήσει που έχουμε λάβει. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε προβλέψει στις 24 και 25 Ιανουαρίου να μας κάνει την παρουσίαση της έκθεσης της η Μαρή Τερέζ. Και θα πρέπει να πάει και στο διαδίκτυο να δει τις απαντήσεις που πήρε η Κομισιόν. Θα τις βρει στην πλατφόρμα της Κομισιόν. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό για να να πει και να προσθέσει την έκθεσή της ορισμένα πράγματα από αυτές τις απαντήσεις. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα άκουσα από τις διάφορες από τις διάφορες παρεμβάσεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε. Αυτός ο κλάδος του πολιτισμού και της δημιουργικότητας τι καλύπτει. Και θα πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε πριν κάνουμε συγκεκριμένε προτάσει. Βέβαια, για το στόχο συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε να δώσουμε μια πρόθεση, να απελευθερώσουμε το δυναμικό του κλάδου. Και ε, τώρα το πρόβλημα είναι τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να απελευθερωθεί, να αποδεσμευτεί αυτό το δυναμικό, για να επιτρέψουμε την ανάπτυξη και την άνθηση αυτών των κλάδων στη νέα ψηφιακή ε, κοινωνία.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 Περιμένουμε την παρουσίαση της έκθεσης. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα, στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Χάνου από τη Φιλανδία. Πόσους Ρωμά έχετε παρεμπιπτόντως εσείς? Um, we're going to have about... Περίπου 5 με 6 χιλιάδες στη Φιλανδία. Στα φιλανδικά τώρα. 5 πάνω πάνω στα φιλανδικά και περίπου όσους και Σάμι. Στην Λαπωνία βέβαια και όχι στην Φιλανδία γενικότερα είναι η Σάμι. Προσπαθώ να είμαι σύντομος, μια που γνωρίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν λάβει το κείμενο και αυτά τα οποία σας λέω α, ήδη τα έχουν μελετήσει. Πάντως πρέπει να ευχαριστήσω τους οικειώδες ηγητές που με βοήθησαν. Θεωρήσαμε ότι θα παγώσει το θέμα των τσιγκάνων. Να που ανέκυψε σήμερα. Και χθες, είχαμε μια δημοσία ακρόαση για τους ε, τσιγκάνους και οπότε τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στη σύνταξη μιας έκθεσης για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πούμε πως εάν θέλουμε να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας, αυτό θα γίνει μέσα από την παιδεία και την εκπαίδευση. Έτσι δίνει τη ευκαιρία σε κάποιο πρόσωπο να έχει τον πρώτο εξοπλισμό, τα μέσα για να προχωρήσει στη ζωή του, να προοδεύσει. Προσπαθούμε να έχουν ίσες ευκαιρίες όλες στη Φιλανδία όσον αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία. Γιατί αν δεν έχουν κάποιες ευκαιρίες δεν υπάρχουν και ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα το, πραγματικό, το ουσιαστικό τώρα είναι να ενθαρρύνουμε τους γονείς τη να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αλλά και οι ίδιοι οι γονείς ενθαρρύνονται να ε, πάνε σε κάποιο σχολείο, σε κάποιο πανεπιστήμιο για να βελτιώσουν το μέλλον τους. Όμως, ο αναφορισμό είναι πάρα πολύ υψηλό για τους τσιγκάνους. Για να ρίξουμε μια μάτια στα στατιστικά όσον αφορά την συμμετοχή στη διαδικασία της ε, παιδείας. Βλέπουμε ότι οι επιδόσεις πάρα πολύ χαμηλές, απουσιασμός, ποικιλία λόγων. Βέβαια, ε, τι περιμένει κανείς, πώς θα πάνε τα παιδιά σχολεία μου, δεν θέλουν να πάνε ούτε οι γονείς. Πολλές φορές θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσκοληθούν στις παραδόσεις τους και να μην πάνε στο σχολείο. Ένας από τους λόγους τους πολλούς είναι και αυτός. Βέβαια, πολλές φορές ο λόγος είναι η φτώχεια. Δεν μπορούν τα παιδιά στο σχολείο, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν παπούτσια να φορέσουν. Επίσης ε, φοβούνται ότι θα είναι αντικείμενα δυσμενής διάκρισης αν πάνε στο σχολείο. Ας κάτσουμε να σκεφτούμε εμείς οι ίδιοι πώς τους φερόμαστε. Παρά τα ωραία λόγια και τα ωραία κείμενα που έχουμε. Μέσα στην καρδιά μας δεν τα πιστεύουμε. Επομένως, θα πρέπει πρώτα εμείς να πιστέψουμε αυτά τα οποία εξαγγέλουμε και να πιστέψουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια σημασία και έτσι να τους εντάξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα Κάπου εδώ θα βάλω τελεία κυρία Πρόεδρε και επί τη βάση των όσων διάβασαν οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες. Μη με παρεξηγήσετε. Δεν ε, δεν το εννοούσα. Σκεφτόμουν κάτι άλλο, μάλλον αφηρημένο. Ναι, ναι, ίσως πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο Τάκουλα ότι το θέμα του σχολείου, του πολιτισμού είναι κέρια σημασίας για να μπορέσει να ενταχθεί ο πληθυσμός των Ρωμά. Άρα χαίρομαι για το γεγονός ότι στις κοινωνίες μας πρέπει ή υπάρχουν ή πρέπει να δημιουργηθούν, θα δούμε, τα ίδια δικαιώματα για όλους. Εάν υπάρχει δικαίωμα, υπάρχει και υποχρέωση συνήθως. Επομένως, υπάρχει υποχρέωση όλων μας για ε, να στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν αυτά που είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα. Αν κάποιος δεν ξέρει να διαβάζει και να γράφει, δεν μπορεί να βρει και δουλειά. Και αν δεν βρει δουλειά, δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια κοινωνία. Σε μια... Και δεν μπορεί να βοηθήσει με ένα υγιή τρόπο να αναπτυχθεί και η κοινωνία. σε όλες ε, τις κοινωνίες μας ε, υπάρχει, αντιμετωπίζουμε προβλήματα για να πείσουμε τους γονείς ε, Ρωμά να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο. Σε μια άλλη επιτροπή σήμερα το πρωί, στην Επιτροπή Ρέτζι, η Κομισιό μας υπενθύμησε ότι πόροι υπάρχουν και υπάρχουν και πολλοί. Αλλά απλώ πολλές φορές τα χρήματα δαπανώνται με λανθασμένο τρόπο σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό θα πρέπει να το μελετήσουμε περαιτέρω και σε όλα τα εργαλεία, αν θέλετε, ένταξης πέραν ε, της, ε, του σχολείου θα έπρεπε να αναφέρουμε και τον αθλητισμό σαν μέσο ένταξης ή ο εθελοντισμός επίσης. Ε, πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να συμμετέχουν κοινωνικά. Ένα άλλο στοιχείο για την κοινωνική ένταξη είναι οι Ρώμα, να θεωρήσουν ότι, τους, ότι είναι προς όφελός τους να αποκτήσουν ένα σπίτι σταθερό. Διότι αν έχουν ένα σπίτι μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στην ε, κοινωνία. Και η κοινωνία δεν θα τους τρέψει ε, τα νότα.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 ε, είναι σημαντικό να λύσουμε το πρόβλημα των Ρωμά που πάνε στο σχολείο. Είναι αλήθεια ότι πολλοί δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο γιατί ο δεν τους υποχρεώνει να κάνουν κάτι τέτοιο ο δικός τους ο νόμος και δική τους η κουλτούρα ή γιατί πράγματι δεν θέλουν να προκαλέσουν την κοινωνία η οποία κοινωνία α, πολλές φορές όπως έχει συμβεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης ε, η ντόπια κοινωνία βγάζει τα παιδιά της από το σχολείο όταν εμφανιστούν τα τσιγκανάκια είναι λοιπόν πρόβλημα αυτό. Επίσης η δική τους κουλτούρα και ο δικός τους νόμος ε, λέει, ότι δεν χρειάζεται να αναγνωρίσουν τις αρχές της χώρας στην οποία τυχαίνει να βρίσκονται ε, ή να ακολουθήσουν τους νόμους της χώρας αυτής. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα μόρφωσης των παιδιών Ρωμά θα πρέπει μοιραία να φτιάξουν ένα πρόγραμμα στο οποίο να συμμετέχουν και οι γονείς και οι γονείς αυτών των παιδιών Βεβαίω. τα εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση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 που, που, χρησιμοποιεί, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα παραδοσιακά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε διότι από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στις χώρες μέλη της ε, Ένωσης τα τσιγκανάκια πάνε σχολείο μοναχά πέντε χρόνια. Αυτό είναι ο μέσος όρος εκπαίδευσης που παίρνουν τα παιδιά αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε δημιουργικοί εδώ εφάνταστοι να πάρουμε, ε, να βρούμε τρόπους να αλλάξουμε τις, ε, τα πρότυπα με τα οποία ζουν οι άνθρωποι αυτοί αν θέλουμε τέλος πάντων να ζουν στις χώρες μας ε, αποδεχόμενοι το δίκαιο των χωρών μας. Επίσης, για να Τελειώνοντας να πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τις ιδιαιτερότητες του κάθε ενός κράτους μέλους που φιλοξενεί η Ρωμά. Γιατί ακριβώς και, και από εκεί και πέρα να κάνουμε και διάκριση μεταξύ των διαφόρων Ρωμά που πάνε στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν πολλές φυλές ε, ε, τσιγκάνων που πηγαίνουν στις διάφορες χώρες για να μπορούμε και εμείς να προσαρμοστούμε και αυτοί να προσαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα της σημασίας της εκπαίδευσης, αλλά πιστεύω ότι, έχουμε, ότι πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Ε, αναφέρθηκε ο φόβος των παιδιών, των γονέων, συγγνώμη. Είναι θέμα πολιτισμικό, πιστεύω. Ε, και, και σε αυτό το τομέα κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή και τον πολιτισμό και το, την κληρονομιά των Ρωμά. Τις αγνο, τα αγνοούμε. Ε, υπάρχει μια αρνητική εικόνα αυτής, ε, αυτών των κοινωνιών. Θυμηθείτε τι έγινε στην, ε, στη χώρα μου φέτος το καλοκαίρι. Πολύ αρνητική εικόνα. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προτάσεις στον τομέα αυτό. Όταν ε, η Μαρία ε, παρουσίασε την έκθεσή της, ε, μιλήσαμε για την κατάρτιση, για την επαγγελματική κατάρτιση και θα πρέπει και πιστεύω να εκμεταλλευτούμε και την, τις πολιτιστικές ικανότητες αυτού του, του λαού. Και αυτό που είπε ο Μάρκο Κορέα είναι πάρα πολύ σωστό. Στις συζητήσεις που είχαμε μετά το φετινό καλοκαίρι, είδαμε ότι αυτό, αυτοί, οι άνθρωποι έχουν, πολλά, έχουν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό το οποίο δεν το χρησιμοποιεί κανείς. Μόλις τώρα έφτασα από την Ουγγαρία. Και εγώ και η Λίβια και είναι πάρα πολύ θετικό Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά αυτή που γίνεται όσον αφορά τους τσιγκάνους. Αυτή η στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική για τους ε, Ρωμά, για τους τσιγκάνους. 6.000 είναι στην Φιλανδία τσιγκάνοι, αλλά στη χώρα μας είναι 500-600.000. Έχουμε τη... Επομένως αυτές τις ε, μειονότητες έχουμε ε, τους καταβλισμούς τους ε, και στη δική μου πόλη που υπάρχουν πολλοί τσιγκάνοι αλλά ζουν σε πάρα πολύ άσχημες συνθήκες νερό, ηλεκτρισμός δεν υπάρχει πάντα οι δουλειές που κάνουν δεν έχουν σχέση με το μέσο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά σε κάθε χώρα άλλα ισχύουν για τους συγκάνους κάθε χώρας, σε άλλη κοινωνική κατάσταση τους διέπει και από πλευράς ένταξης κοινωνικής, από πλευράς πολιτισμού, πολλάς, παιδε, παιδείας και αυτά είναι πολύ σημαντικά, να ληφθεί όμως υπόψη και ο οικονομικός παράγον. Ε, άμα πεινάνε τα παιδιά σε μια ε, οικογένεια, τι να τους πούμε για κουλτούρα, για πολιτισμό. Θα πρέπει οι βασικές ανάγκες να έχουν καλυφθεί. Ε, σας λέω τι γίνεται σε Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και μέσω του αθλητισμού μπορεί να γίνει η ένταξη κοινωνική. Φυσικά είναι αλληλένδετη η κοινωνική ένταξη με την οικονομική ένταξη. Το ένα οδηγεί στο άλλο. Πάντως πάρα πολλοί από τους τσιγκάνους δεν αναγνωρίζουν την κρατική εξουσία όπως ε, προαναφέρθηκε. Πάντως, εγώ έχω πάρα πολύ θετικές εμπειρίες από ε, τη δουλειά μας με τους τσιγκάνους, όμως υπάρχουν ε, πάρα πολλές προκαταλήψεις εναντίον τους, Πολλέ αρνητικέ προκαταλήψεις. Το κράτο θα πρέπει να είναι ο φύλακα των δικαιωμάτων των τσιγκάνων και συνάδελφοι είναι πάρα πολύ βασικό να σα πω το εξή ότι εμεί εδώ ω ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω θεσμικό όργανο, ερετό, εκλεμμένους πολίτε, έχουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ότι δηλαδή θα πρέπει να εντοπίσουμε όλα αυτά τα ακροδεξιά κόμματα τα οποία ε, βάλουν κατά των ε, τσιγκάνων και αυτό να τον ληφθεί υπόψη για τη μελλοντική μας στρατηγική, πολιτική, να καταπολεμήσουμε αυτές τις ε, πολιτικές ομάδες που θέλουν να τους αποστερήσουν από δικαιώματα. πολιτισμός, παιδεία είναι πολύ σημαντικά. Και από την άλλη μεριά, οικονομικός παράγον. Επομένως και για άλλη μια φορά και πάλι σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στο, στο έργο του δικό μου και της συναδέλφου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι η πρόταση του συναδέλφου μας υπάρχει μόνο στα αγγλικά, αλλά μέχρι τις 18 Δεκέμβρη θα έχουν γίνει όλες οι μεταφράσεις. Και τότε μπορείτε να καταθέσετε και τις απολογίες σας. Αυτά το έχετε διαβάσει. Θα ήθελα να ζητήσω ε, συγγνώμη από τον κύριο Τάκουλα, γιατί δεν ήμουν εδώ για να ακούσω την παρέμβασή του, αλλά άκουσα σε γενικές γραμμές ε, ε τις, τις προτάσεις του χτες στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Θα ήθελα να προσέξουμε κάποια πράγματα ε, από αυτά που άκουσα τουλάχιστον δεν θα πρέπει να προβάλλουμε τα ίδια στερεότυπα απέναντι στην κοινωνία των Ρωμά. Θα πρέπει να μην τους, ε, επιβα... να μην ε, τους βλέπουμε με με κάποια στερεότυπα, π.χ. ας πούμε, ότι οι, οι Ρωμά είναι εγκληματίες. Όντως, μπορεί να υπάρχουν εγκληματικά στοιχεία, αλλά το το, αυτή τη στιγμή εξατομικεύουμε τις ποινές και δεν θα κατηγορήσουμε συλλήβδιν μια ολόκληρη κοινωνία. Τώρα, επίσης τίθεται το θέμα τι σημαίνει πολιτιστική διαφοροποίηση, τι σημαίνει σεβασμός της πολιτιστικής διαφοροποίησης, διότι το να σεβαστούμε την πολιτιστική διαφοροποίηση δεν είναι να τους βάλουμε όλους στο ίδιο καλούπι. Και εγώ πιστεύω ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής δια... διαφοροποίησης δεν είναι να τους βάλουμε σε ένα καλούπι, είναι, δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε την αφομοίωση με την ένταξη. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, στη συζήτηση είναι ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα της κοινωνίας των Ρώμα αυτή τη στιγμή. Ένα, μεγαλύτερο, ένα μεγάλο μέρος του ε, πληθυσμού εγκαθίσταται μόνιμα κάπου πλέον και το κάνει αυτό για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Επομένως θα πρέπει να σταματήσουμε με αυτά τα κλισέ που λένε ότι οι τσιγκάνοι, οι Ρωμά δεν θέλουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ίσα ίσα έχουμε πολύ καλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι μπορούν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο και πηγαίνουν στο σχολείο. Τώρα γιατί δεν πηγαίνουν αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Και όταν το κάνουμε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι η διακρι... ποια είναι η διακριτική μεταχείριση ε, που υφίστανται τα παιδιά αυτά. Όταν δηλαδή, είχα πάει στη Ρουμανία, είχα συζητήσει με διάφορους Ρωμά, ε, Ρουμάν, ήταν Ρουμάνοι και κάνανε διάφορες, πηγαίνουν έρχονταν ανάμεσα στη Ρουμανία και στη Γαλλία, διότι θέλαν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στην σχολείο στη Γαλλία, γιατί στη Γαλλία αισθανόντουσαν πιο ήσυχοι, πιο ασφαλείς. Λοιπόν, αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, γιατί αλλιώ δεν θα το δούμε το, το πρόβλημα στις σωστέ του διαστάσεις. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα κλισέ κυρίως. Πρέπει να πω ότι η έκθεση αυτή με, με βρίσκει σύμφωνη. Αλλά καταρχάς θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα καλά παραδείγματα σχολικής ένταξης μέσω των εμπειριών που έχουμε, είτε θετικών είτε αρνητικών, ένα τρόπο για να ξεπεράσουμε τα κλισέ είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τους Ρωμά. Ε, να δούμε τι καλές εμπειρίε ε, ένταξη. Και θα το δούμε σε διάφορε επιτροπές. Δεύτερον, συμφωνώ με συνάδελφο με τη συνάδελφο που είπε ότι η μόνιμη εγκατάσταση των Ρωμά είναι, γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι φανταζόμαστε ενδεχόμενα. Οι καταβλισμοί και ο νομαδισμός δεν αφορά το σύνολο της κοινότητας των Ρωμά. Μιλάμε για άτομα τα οποία είναι πρόσφυγες, τα οποία είναι παράνομοι μετανάστες, ε, μπορεί να έφυγαν από κάποιες περιοχές όπου υπήρχαν διενέξεις κτλ. Βέβαια θα πρέπει και ακόμα και στους καταβλισμούς να έχουμε κάποιες δυνατότητες, διότι αλλιώς τα παιδιά αυτά δεν θα μπορούν να πάνε ποτέ σχολείο και για, την, ε, τη χώρα μου έχω στο μυαλό μου το Τρέντο που είναι μια συγκεκριμένη πόλη, μια ιδιαίτερη πόλη. Τρίτο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εργαστούμε με τις οικογένειες και το έχω δει αυτό. Συμφωνώ με τον Ιβάν όταν το έλεγε αυτό. Είχα την... Ε, εγώ είχα την εμπειρία ε, ηγέτες, ε, από ηγέτες των, της κοινότητας των Ρωμά που λέγανε ότι θέλουν να στείλουν τα παιδιά σχολείο αλλά δεν υπήρχαν τα απαραίτητα, οι δεν υπήρχαν χρήματα θα πρέπει να δώσουμε και κάποια κίνητρα, πιστεύω. Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και αντικίνητρα. Γιατί αυτή τη στιγμή πέραν της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν είναι πολλά τα παιδιά που προχωρούν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώ στον συγητή και πάλι το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι το θέμα της ενσωμάτωσης των Ρωμά δεν ε, είναι μοναχά πολιτιστικό. Δεν έχει μοναχά την πολιτιστική πτυχή την οποία συζητούμε εμείς εδώ σήμερα και την πτυχή της εκπαίδευσης υπάρχουν και άλλες πτυχές οικονομικές και άλλες της ενσωμάτωσης των Ρωμά. Γενικότερα η κατάσταση των Ρωμά σε διάφορες χώρες είναι διαφορετική και η κατάσταση στην Ουγγαρία και στην Ρουμανία παραδείγματο χάρη είναι τελείως διαφορετική από την κατάσταση των Ρώμα στη Φινλανδία. Στην, ε, η ενσωμάτωση των Ρώμα στη Φινλανδία είναι ε, πάρα πολύ επιτυχής. Εγώ στο Πανεπιστήμιο είχα συμφοιτητές Ρώμα, φίλους Ρώμα, άρα η κατάστασή τους στη Φινλανδία και η ενσωμάτωσή τους είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες χώρες. Δεν άκουσα Βεβαίω δεν άκουσα εδώ κανένα από τους ομιλητέ που μίλησαν για να μιλήσω για το στίγμα που φαίνεται να υπάρχει για τους ο, ο, ε, δεν, κανείς δεν θέλει να στιγματίσει τους ο, τσιγκάνους εδώ στην, ε, στις Βρεξέλλες, στην Ευρώπη, την πολιτισμένη Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα και εμείς οι οποίοι έχουμε τα μέσα θα μπορούσαμε ίσως να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω αυτούς που είναι σχεδόν αποκλεισμένοι από την κοινωνία μας. Όπως έχουμε και εμείς μια ζωή, έχουν και αυτοί. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω γιατί δεν θέλω να κάνω κήρυγμα και να με κατηγορήσετε μετά ότι κάνω κηρύγματα, λέ, ε, κλείνω λέγοντας ότι περιμένω τις τροπολογίες σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Λοιπόν, στις 8, όχι στις 18 Δεκεμβρίου, θα είναι έτοιμες οι μεταφράσεις και από εκεί και πέρα μπορείτε να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Συγγνώμη, έκανα λάθος λέει η πρόεδρος. Μίλαγα για την άλλη γνωμοδότηση του Χάνου. 15 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών. Εντάξει. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. Θα ήθελα να ζητήσω από αυτούς που δεν είναι συντονιστές να φύγουν από την αίθουσα. Μένουμε εδώ μόνο οι συντονιστές. Ε, ποιος μείνει από τους σοσιαλιστές, Μαρία.